Uh, So good afternoon, ladies and gentlemen. Um, If uh, I could invite you to find a seat. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ καθίστε. Καλώς ήρθατε στη σημερινή μας απογευματινή ακρόαση. Welcome also to anybody who's watching. Και καλώς ήρθατε σε όσους μας παρακολουθούν ε, στο διαδίκτυο. ειδικότερα αν συμμετέχετε σε ηλεκτρονική επίλυση διαφορών ή στην εργασία επί του θέματος αυτού, θα θεωρήσετε την ακρόαση αυτή πολύ σημαντική και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης πολύ σημαντική. Θα ήθελα να σας πω ορισμένα πράγματα για το πρόγραμμά μας σήμερα το απόγευμα. Δύο ώρες έχουμε στη διάθεσή μας για την ακρόαση. Θα δώσω το λόγο σε λίγο στους δύο εισηγητές της Επιτροπής μας, που είναι επικεφαλής των εργασιών μας σε δύο πολύ σημαντικές ε, νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής ε, για τον Επίτροπο των Καταναλωτών, ε, τον κύριο Ντάλι, έχουμε τον κύριο Γκρέκ, ο οποίος θα μας μιλήσει για την εναλλακτική πύληση διαφορών και έχουμε ε, την ε, κυρία Τουν, η οποία ε, θα είναι υπεύθυνη, θα μας παρουσιάσει την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών. Θα ήθελα να καλωσορίσω και την εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ που θα πάρει και εκείνη το λόγο κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι επειδή είναι εδώ μαζί μας ε, εμπειρογνώμονες, τους οποίους βέβαια θα παρουσιάσω ε, και στη συνέχεια, Ούρσουλα Πακ από την ΠΕΟΚ, ο κύριος Ολιβιέρα από την Business Europe, ε, ο Δόκτωρ Παύλο Κορτές από το University του Λέστερ και η Καταζίνα Λαζότα από την Εντίμα. Θα σας πω μερικά πράγματα περισσότερα για τους ομιλητές μας όταν θα τους παρουσιάσω για να λάβουν το λόγο. Ε, έχουμε επίσης τον κύριο Πεγκάτολης, ο οποίος δεν ξέρω πού είναι. Ανάτος. Ναι, ναι, τώρα σας βλέπω. Καλώς ήρθατε που ήταν ε, ο εισηγητής ε, για την η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και αν θέλει κάποια στιγμή να πάρει το λόγο, ευχαρίστως. Αυτά λοιπόν έχουμε μπροστά μας, δύο ώρες έχουμε στη διάθεσή μα και θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον Λουί Γκρέκ για να μας κάνει κάποια εναρκτήρια σχόλια και μετά θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Τουν και μετά στου ομιλητές μας. Λουί, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι παρά το γεγονό ότι υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ απόψει για ε, πολύ ειδικά ζητήματα, νομίζω ότι σε γενικέ γραμμέ μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει ανάγκη νομοθετική ε, ε πρόταση για την ε, εναλλακτική επίλυση διαφορών. Όταν τη γνωρίζουν, ε, ε, οι καταναλωτές θεωρούν ότι οι ποιοτικέ ιδέες λειτουργούν. Σύμφωνα με, το 2010, ε, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2010, πολύ λίγοι καταναλωτές υπέβαλαν καταγγελίες στην εναλλακτική επίλυση διαφορών. Δεν ε, συμμετέχουν εύκολα οι καταναλωτές ε, σε αγορές διαστηνοριακές ε, μέσω του ίντερνετ. Πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι το εξίσου υψηλό το επίπεδο προστασίας, είναι μεγάλη σημασία κατά την άποψή μου η οδηγία να μην αφορά μόνο τις διασυνοριακές διαφορές, αλλά και εντός ενός κράτους μέλους ε, γιατί διαφορετικά ε, δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της άνησης μεταχείρισης του Σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να έχουμε ένα ισότιμο επίπεδο ε, αποτελεσματικότητας και προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Όσον αφορά τώρα τον προσανατολισμό, η ηλεκτρονική επίλυση διαφορών πρέπει να είναι απλή, γρήγορη, όχι πολύ γραφειοκρατική και οικονομική. Πρέπει δηλαδή να έχει, κάποιες, ε, να έχει κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με τις, ε, τους συμβατικούς τρόπους επίλυσης ε, διαφορών. Κατά την άποψή μου πρέπει να ενθαρρύνουμε τη χρήση ε, συστημάτων διαχείρισης ώστε τα προβλήματα των καταναλωτών να μπορούν να λυθούν με το συντομότερο δυνατό τρόπο και να μην υπάρχει λόγος πάντοτε να καταλήγουμε σε έναν φορέα ADR, δηλαδή ε, εναλλακτική επίλυση διαφορό. Πρώτα θα θέλουμε να έρθουν σε επαφή με τον έμπορο πριν ε, απευθυνθούν στον φορέα αυτό. Εγώ ε, είμαι υπέρ της ελάχιστης εναρμόνισης, ε, γιατί όπως αναφέρεται και στην αξιολόγηση δικτύπου της Επιτροπής, ε, θα ε, σημαίνει ότι θα συμμετέχουν περισσότεροι παίκτε. Επίση, τα κράτη-μέλη πρέπει να μπορούν να είναι ελεύθερα να επιλέξουν υψηλότερα επίπεδα ε, προδιαγραφών από αυτά που προτείνει η ε, οδηγία. Εμείς θέλουμε μια εναρμόνιση ελάχιστη, εναλλακτικές προσεγγίσεις, εναλλακτική επίλυση διαφορών, ενώ παράλληλα εγκαθιδρύουμε ένα συγκεκριμένο σύνολο προτύπων όταν εφαρμόζεται σωστά η οδηγία, ο καταναλωτής πρέπει να έχει πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου αμερόληπτη, ε, μηχανισμό αποζημίωσης και επίλυσης ε, της διαφοράς που τον απασχολεί από απόψεως αποτελεσματικότητας. Η, πρόταση η οποία δεν, ε, είναι, δεν καθιστά υποχρεωτική την ε, επίλυση μέσω ADR διατηρεί τις, ε, τους υπάρχοντες φορείς ε, ADR σε, στο βαθμό βέβαια που λειτουργούν αποτελεσματικά. Εγώ εκ πρώτης όψεως συμφωνώ ε, με το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής αλλά αναγνωρίζω την ανάγκη μιας πρακτικής προσέγγισης και επέκτασης ειδικότερα για περιπτώσεις που είναι πολύ τεχνικές ή πολύ περίπλοκες. Οι διαδικασίες ADR πρέπει να είναι ε, είτε δωρεάν είτε ε, πολύ μικρού κόστους. Ε, το, να το επιτύχουμε αυτό θα σημαίνει ότι είναι ελκυστική διαδικασία για τους καταναλωτές γιατί συχνά απογοητεύονται από το υψηλό κόστος των, της διαδικασίας επίλυσης διαφορών. Η πρόσβαση στις πληροφορίες επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Για το Solvit, για παράδειγμα, είναι μια ε, πρωτοβουλία η οποία δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες γιατί υπήρχαν, υπήρχε πολύ χαμηλό ποσοστό ευαισθητοποίησης από πλευράς καταναλωτών. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες ε, είναι ακριβείς, ανεξάρτητες, ε, προσπελάσιμες και φιλικές προς τον καταναλωτή και πρέπει να ε, εξασφαλίζουμε ότι είναι πρακτικές οι πληροφορίες και αποτελεσματικές και οικονομικές. Τα κράτη-μέλη πρέπει επίσης να αναλάβουν τον δικό τους ρόλο και να εξασφαλίζουν ότι οι φορείς ADR ε, είναι αποτελεσματικοί με παρακολούθηση της ε, αποδοτικότητάς τους. Ε, ζητήματα ελευθερίας πρέπει να ε, τα εξετάσουμε επίση και θα ήθελα να ζητήσω κατευθυντήριε γραμμές από την Επιτροπή ε, για έναν κώδικα συμπεριφοράς, ε, παρακολούθηση, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και διάδοση πληροφοριών μεταξύ των φορέων ADR. Επιπλέον, κατά την άποψή μου, όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι εκπρόσωποι τους πρέπει να παίξουν ένα ρόλο στη διαδικασία, ώστε να υπάρχει ευρύτερη συνένεση, ισορροπία και υποστήριξη για την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Θέλουμε ένα σύστημα ε, λογοδοσίας, διαφανές, ε, δεν θα πρέπει να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και θα έπρεπε να καταλήγει σε μία απόφαση που να είναι δίκαιη και ανεξάρτητη. Υψηλό επίπεδο διαφάνειας θα βελτιώσει την αξιοπιστία ενός συστήματος ADR μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, αλλά επίσης θα παρέχει δεδομένα που θα βοηθήσουν ε, στην ε, ε, βελτίωση συνεχώς των φορέων αυτών με την ADR στο πλαίσιο μιας ενιαίας αγοράς βασικό θέμα είναι η εμπιστοσύνη. Αν οι καταναλωτές ε, εμπιστεύονται τους φορείς αυτούς και αν διαπιστώσουν ότι δουλεύει καλά και για τα δύο μέρη θα αρχίσει η εφαρμογή του μηχανισμού αμέσως και έτσι μπορούμε να ενισχύσουμε την ενιαία αγορά, ειδικότερα την ψηφιακή αγορά, η οποία θα είναι υποφελής για την ευρωπαϊκή κοινωνία και θα βοηθήσει στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη. Στα Ιταλικά λέμε ότι το καλύτερο είναι ο ε, εχθρός του καλού. Είναι πολύ καλή η ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ε, πρέπει να βελτιωθεί. Έχουμε μια καλή βάση, αλλά αν επιμένουμε και θέλουμε να πετύχουμε την τελειότητα, δεν θα έχουμε καθόλου ε, αποτελεσματική ε, και χρήσιμη οδηγία στο τέλο. Οπότε πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε τι βελτιώσει, αλλά πρέπει να καταλήξουμε και σε μια οδηγία που θα βοηθήσει του έμπορου και του καταναλωτέ πολύ σύντομα. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, και τώρα, κυρία Τούν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λουί Γκρέχ, διαβάζοντας αυτά τα έγγραφα, Λυπάσω ότι δεν είναι ένα έγγραφο και μοναδικό, αλλά δύο. Και τα δύο έγγραφα είναι αλληλένδετα, ή θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον. Και θέλουμε να συνεργαστούμε στενά επί των δύο εγγράφων. Διότι η, δια... η διευθέτηση διαφορών στο διαδίκτυο είναι το να δημιουργήσει εμπιστοσύνη, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη όσον αφορά το εμπόριο στο διαδίκτυο, κυρίω σε δυσυνοριακό επίπεδο. Είναι μεγάλο το διακύβευμα. Θα είδατε πρόσφατα την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί δείχνει ότι η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ενίας Αγοράς, της ψηφιακής Ενίας Αγοράς, θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κατά 110 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μέχρι τόσο και όλα εξαρτώνται κατά πολύ από την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ε, προς την ψηφιακή αγορά. Για να τονωθεί το διασυνοριακό διαδικτυακό εμπόριο ε, χρειάζονται πολλά στοιχεία να ληφθούν υπόψη και μπορούσαν να μας βοηθήσουν να προωθήσουμε το διασυνοριακό διαδικτυακό εμπόριο. Βλέποντας το όλο σκηνικό το ευρωπαϊκό, βλέπει ότι δύο στα τρία ευρωπαϊκά νοικοκυριά έχουν σύνδεση με το διαδίκτυο, αλλά μόνο 12% χρήστε του διαδικτύου αισθάνονται ότι είναι ασφαλεί για να κάνουν αγορέ ε, σε διαδικτυακό επίπεδο. Όλοι ξέρετε του αριθμού. Απλώ ήθελα να σα του θυμίσω εκ νέου. Ένα τρίτο των καταναλωτών θα θεωρούσε την αγορά στο διαδίκτυο από άλλη χώρα, γιατί βρίσκει κάτι φθηνότερο ή καλύτερο προϊόν αλλά μόνο 8% κάνουν πράγματι, πραγματοποιούν την αγορά. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι ένα σύστημα το οποίο είναι εύκολο, διαφανές, φιλικό προς το χρήστη, που δίνει το, την εντύπωση, το συνέστημα στον καταναλωτή να είναι ασφαλέστερος. Ο, ότι το μέσο αυτό πραγματικά τους βοηθάει και δεν χάνονται στο διαδίκτυο. Αυτό προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν συνέταξε μάλιστα αυτό το έγγραφο για την ε, διαδικτυακή επίλυση των διαφορών. Πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει. Αυτή τη διαδικτυακή επίλυση των διαφορών θα έπρεπε να είναι ένα σύστημα στο οποίο μπορεί να αποστέλλονται μηνύματα διαδικτυακά, να μπορεί να απευθυνθεί σε μια ιστοσελίδα όταν έχει πρόβλημα. Πίσω από την ιστοσελίδα κρύβεται μια βάση δεδομένων. Με όλα τα συστήματα εναλλακτική επίλυση διαφορών, ADR, όλα τα συστήματα που είναι προσβάσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το, τη βάση δεδομένων θα πρέπει να τη συντηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτός που διαμαρτύρεται θα πρέπει καταρχήν να προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβλημα με τον έμπορο πρώτα απ' όλα. Και μόνο όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται για διάφορους λόγους, για γλωσσικούς λόγους, για λόγω παρεξηγήσεων, λόγω μεγάλης γεωγραφικής αποστάσεως. Αν δεν βρίσκεται λύση διμερός, τότε μπορεί ο πολίτης να καταφύγει σε αυτό το εργαλείο, το διαδικτυακό, για να βρει ε, την καλύτερη εναλλακτική λύση επίλυσης διαφορών, τον καλύτερο φορέα εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών που τον βοηθήσει με το πρόβλημά του. Είναι σημαντικότατο το ότι ο διαμαρτυρόμενος αυτός άνθρωπος θα πρέπει να βρει ε, μια δυνατότητα να εκφράσει το, τη διαμαρτυρία του στη γλώσσα που χρησιμοποιεί καλά, τη μητρική του ή άλλη γλώσσα που γνωρίζει καλά. Και έτσι θα του προταθεί του πελάτη διάφορους φορείς επίλυσης διαφορών που μπορεί να καλύψει τον τομέα του, της καταγγελίας του. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση, όμως κατά την άποψή μου υπάρχουν αρκετές ασάφειες θα ήθελα να τη συζητήσω μαζί σας. Ήδη συζήτησα με διάφορους ανθρώπους και με διάφορα κοινοτικά όργανα. Η πρώτη ασάφεια. Μιλάμε για συνοριακό εμπόριο. Τι σημαίνει διασυνοριακό στην ενιαία αγορά και στο διαδικτυακό εμπόριο. είναι κάτι που θεωρώ σημαντικότατο και περιπλοκότατο στο έγγραφο. Όταν είμαστε δεδεμένοι με το διαδίκτυο και στην ενιαία αγορά, δημιουργούνται πολλές καταστάσεις όπου δεν γνωρίζει κανείς από πού αγόρασε. Και δεν γνωρίζει αν η συναλλαγή είναι διασυνοριακή ή όχι, γιατί μετακινήθηκε από τη μια χώρα στην άλλη αφού έκανε την αγορά. Υπάρχουν διάφορε εξαιρέσει. Η πρώτη σαφια αυτή αυτό το σύστημα ADR θα πρέπει να ασχολείται μόνο με διασυνοριακό εμπόριο ή γενικά με το εμπόριο στο διαδίκτυο. Δεύτερη εσάφεια. Είναι αρκετά ολοκληρωμένο το σύστημα. Συνδέεται με όλα τα δίκτυα και τα συστήματα που έχουμε. Μήπως δημιουργούμε και άλλη μια ενιαία θηρίδα πρόσθετη. Μήπως θα μπορούσε να ενταχθεί στα ήδη υπάρχοντα. Έχουμε την, ε, την πύλη, την ηλεκτρονική Europortal που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την επίλυση αυτών των προβλημάτων ή που αποτελεί σημείο επαφής εκείνων που θέλουν να βρουν ένα μηχανισμό επίλυσης διαφορών και διάφορα άλλα δίκτυα θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα στους καταναλωτές. Κάποιοι συναδελφοί μου και οι συγητέ είπαν ότι είναι παραπλανητική ονομασία, διότι NDR είναι, αν θέλετε, ένα σημείο επαφή. Δεν επιλύει τι διαφορέ. σω η διαδικτυακή επίλυση διαφορών είναι παραπλανητική η έκφραση. Αυτό που μα λείπει, μου λείπει εμένα από το έγγραφο, που αλέω είναι πολύ ενδιαφέρον και δημιουργικό, είναι τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών που διευκολύνουν την επαφή του καταναλωτού με τους διάφορους αρμοδίους. Τι ρόλο παίζουν. Και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε εκ νέου. Γι' αυτό ζήτησα δύο έγγραφα ενημερωτικά. Ένα με τα υπέρ και τα κατά της διάκρισης που γίνεται. Θέλουμε διάκριση μεταξύ της διαδικτυακής, μεταξύ διασυνοριακής και μη διασυνοριακής διαδικτυακής επίλυσης διαφορών. Δεύτερον, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα που λειτουργεί αποτελεσματικά. Συνεργαζόμενοι με άλλες ιστοσελίδες Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Συμφωνώ πλήρως με τον κύριο Γκρέκ, τον άλλο εισηγητή. Αυτό που χρειαζόμαστε πραγματικά για να τονώσουμε την ενιαία αγορά είναι να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη στους καταναλωτές. Να έχει εμπιστοσύνη ο καταναλωτή στον έμπορο. Και αντιστρόφω. Να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη. Αυτό είναι άκρο ανάγκαιο και ελπίζω όλα αυτά να τα καταφέρω με μέσω των εργασιών που μόλι ξεκίνησαν πάνω στο θέμα. Καλώ. ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ, διότι μας παρουσιάσατε τους διάφορους τομείς που θέλετε να εξεταστούν από πλευράς προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο χρονοδιάγραμμά μας θα αναφερθούμε στο τέλος της ακροάσεως. Είναι η αρχή της διαδικασίας αυτή. Η ιδεώδης ευκαιρία η Επιτροπή μας να συλλέξει πληροφορίες και να τις διαβιβάσει στους εισηγητές για να τις λάβουν υπόψη σε τυχόν τροπολογίες. Θα ακούσουμε τους φιλοξενούμενους μας που είναι εμπειρογνώμονες και ενδιαφέρονται για τον τομέα θα προσκληθούν να μιλήσουν για 8 λεπτά ο καθένας. Θα έχουμε το ακριβές χρονόμετρό μας, θα τους βοηθά να κρατήσουν το χρονικό τους όριο. Καλωσορίζω τακτικό επισκέπτη μας, πασίγνωστο του Κοινοβούλιο, τον κύριο Πάκτου, την Ούρσουλα Πάκελ, η υποδιευθύντρια του Μπίοκ, γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα πολιτικής καταναλωτών και δραστηριοτήτων καταναλωτών είναι νομικός, ενδιαφέρεται ιδιαίτερο για το θέμα. Ούρσουλα λοιπόν, ας ξεκινήσεις τις παρουσιάσεις των προσκεκλημένων. Έχεις και κάποιες διαφάνειες να μας δείξεις. Λοιπόν, Ούρσουλα πάκε το λόγο, σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ για την... Ευχαριστώ για την ευγενική εισαγωγή σας. Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ που καλέσατε την Μπιούκ σε αυτό το σημαντικό γεγονός. Θέλω να υπογραμμίσω ευθύς εξ αρχής ότι δύο δεκάδες τώρα εκπροσωπούν οι ενώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης των καταναλωτών και ζητούν αυτό το σύστημα. Όλοι ξέρουμε πολύ καλά ότι για τους καταναλωτές είναι πολύ δύσκολο να καταφύγουν στα δικαστήρια. Χρειάζονται μεταξύ άλλων εναλλακτικά μέσα για να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και είμαστε πεισμένοι ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν να το κάνουν και θα είναι ορόσημο στην ιστορία της πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και του δικαίου προστασίας των καταναλωτών. Θέλω να δραθώ τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής γιατί πάντα υποστήριζαν αυτό το αίτημα και πραγματικά απευθύνω έκκληση σε εσά να δραχθείτε τις ευκαιρία να διασφαλίσετε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά με αυτή την ευκαιρία. Είναι μια μοναδική ευκαιρία που έχουμε να τα καταφέρουμε. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί στην νομοθεσία που θα συντάξουμε. Νομοθεσία που όπως επεξηγήθηκε από τον προλαλήσαντα κύριο Γκρέκ θα μπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Η Μπιουκο καλωσορίζει τι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα θα επικεντρωθώ στον περιορισμένο χρόνο που έχω σε λίγα σημεία που πιστεύουμε ότι είναι κλειδιά και έχουν σημασία και πρέπει να παραμείνουν και να διατηρηθούν σε κάποια, και κάποια σημεία που θα σας ζητούσα να βελτιώσετε τα πράγματα ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στις διατάξεις που θα συντάσσονται. Πρώτα απ' όλα για το ADR, για τον προτινόμενο κανονισμό ADR, εναλλακτικών αυτών ε, μεθόδων ε, επίλυσης διαφορών. Υπάρχει εδώ ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και σωστό είναι αυτό να είναι ευρύ, διότι η ίδια φύση του ADR καθώς και το ευρύ φάσμα πρακτικών στην Ευρώπη απαιτούν ένα τέτοιο ευρύ ορισμό και φάσμα. Από την άλλη πλευρά η ανάγκη να να εντάξουμε πολλές τέτοιες ε, προσεγγίσεις δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε χαμηλές προδιαγραφές. Χρειαζόμαστε αναβαθμισμένες υψηλής ποιότητας προδιαγραφές στο ADR. Αλλιώς δεν θα υπάρξει εμπιστοσύνη σε αυτό το σύστημα και δεν θα καταφέρει ο κανονισμός αυτός να είναι επιτυχής και αποτελεσματικός. Φυσικά έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η δημιουργία του ADR συνεπάγεται κόστη είτε για τα κράτη-μέλη είτε για τις επιχειρήσεις. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό για αυτούς τους λόγους είναι να στοχεύσουμε και να επιτύχουμε υψηλές προδιαγραφές φές και ρυθμίσεις, γιατί αλλιώς δεν θα είναι χρήσιμες ή χρήσιμοι. Και υποστηρίζουμε ιδιαίτερα την πρόταση να καλύπτει το ADR σε ένα ευρύ φάσμα. Θα πρέπει να εφαρμόζεται, και αυτό είναι σημαντικό, και στις εθνικές αλλά και στις διασυνοριακές, διακρατικές τέτοιες διαφορές. Και θα πρέπει και τομεακά να είναι ευρύ το φάσμα, όσο το δυνατόν ευρύτερο. Απευθύνουμε έκκληση πραγματικά σε εσά στην Ευρωβουλή να διατηρήσετε αυτά τα στοιχεία στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερα τρία σημεία θα ήθελα να αναφέρω, που δεν μα ικανοποιούν απόλυτα και θα θα ζητούσαμε να τα βελτιώσετε αν γίνεται. Αφορούν κυρίως αρχές που θα θέλαμε εμείς στην πρόταση αυτή να τις εντάξετε. Πρώτα την αρχή της ανεξαρτησίας. Όπως μπορεί να γνωρίζετε η σύσταση για συστήματα ADR του 1998 συμπεριλάμβανε την αρχή της ανεξαρτησίας ως έναν από τους κύριους πυλώνες των συστημάτων ADR. στην νέα όμως πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή η απέτηση απουσιάζει και ανησυχούμε πάρα πολύ για την αφαίρεση αυτής της απέτηση ανεξαρτησίας διότι είναι πραγματικά ένα θεμελιώδες στοιχείο για την εμπιστοσύνη, ώστε να είναι απόλυτα ανεξάρτητο το σώμα, ο φορέας ADR. Και αναγνωρίσουμε στην θετική πλευρά των πραγμάτων ότι προβλέπει την αμεροληψία και αντικειμενικότητα η πρόταση αυτή ως στοιχεία. Αλλά ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα και αμεροληψία δεν είναι τα ίδια πράγματα. Πρέπει να πετύχουμε και την ανεξαρτησία. Σε αυτό το πλαίσιο είναι απόλυτα σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό να θίξουμε το θέμα της, ε, των προγραμμάτων αντιμετώπισης ε, προσφυγών ή παραπώνων ε, όσον αφορά εθνικούς συνδέσμους και υπεύθυνου, που αποκλειστικά θα πρέπει να έχουν αυτό το στόχο μπορούμε να κατανοήσουμε ότι μπορεί να υπάρχει πίεση από τις επιχειρήσεις ε, να ε, διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο να διαμορφωθούν με αυτόν τον τρόπο τα πλαίσια της ε, οδηγίας για την επίλυση με προγράμματα, για προγράμματα επίλυσης διαφορών. Όμως θα πρέπει να προσέξουμε, διότι στο παρελθόν γνωρίζουμε από την ίδια την πείρα των αδελφών οργανισμών ότι τέτοιου είδους προγράμματα <clears throat> παρουσιάστηκαν στους καταναλωτές ως ανεξάρτητα προγράμματα, ενώ στο τέλος τέλος λειτουργούσαν μόνο υπέρ των επιχειρήσεων. Αυτό λοιπόν πάλι υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και δεν οδηγεί τους καταναλωτές να στρέφονται στην χρήση ή στην προσφυγή του ADR. Είναι κέρια σημασία οι στο άρθρο 2 της προτινόμενης οδηγίας να είναι απόλυτα σαφής και οι διατάξεις για την εσωτερική επίλυση, εναλλακτική επίλυση διαφορών να μην ε, έχουν τέτοια περιθώρια ώστε να παρεκκλίνουν ε, σε κάποιους που δεν θα πρέπει να εντάσσονται στην ADR. Σε σχέση με την δεύτερη σημαντική αρχή που δεν εντάσσεται μέχρι σήμερα σε αυτή την προτινόμενη ε, οδηγία είναι η αρχή της νομιμότητας και θα ήθελα εδώ να υπεξηγήσω κάτι, να καταστήσω απόλυτα σαφές ότι η αρχή της νομιμότητα είχε ενταθεί στην προηγούμενη ρύθμιση. Ουσιαστικά τι σημαίνει με απλά λόγια, να το πω έτσι, ότι ο καταναλωτή δεν μπορεί να, <clears throat> αφαιρε, να των δικαιωμάτων και των διατάξεων που ισχύουν στη χώρα του. Και από το παρελθόν κιόλα. Θέλουμε αυτή η αρχή που οι ενώσει καταναλωτών θεωρούν ότι είναι σημαντικότατο για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών πρέπει να παραμείνει. Είναι σημαντικό για τι ε, κρατικέ εθνικέ υποθέσει να μην βρεθούν οι καταναλωτέ μέσω μια απόφαση ADR σε χειρότερο υποβαθμισμένο επίπεδο ε, σε σχέση με το τι θα συνέβαινε μέσω της προσφυγής δικαστηρί, σε δικαστήριο. Όμως είναι σημαντικό και διασυνοριακά, όπου θα πρέπει να είναι βέβαιοι οι καταναλωτές ότι δεν θα βρεθούν σε ένα υποδέστερο επίπεδο σε σχέση με εκείνο που θα ίσχυε στη χώρα τους. Θέλουμε λοιπόν να σας ζητήσουμε να επαναενταχθεί αυτή η αρχή της νομιμότητας και θέλουμε να αναφέρουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο και πάλι ότι η Ευρωβουλή και ιδιαίτερα η δική σα Κοινοβουλευτική Επιτροπή μεγάλο έργο επετέλεσε για την οδηγία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την προσέγγιση των αρχών ε, σε σχέση με θεμελιώδεις αρχές δικαίου και σημειώθηκε πρόοδος και πρέπει να διευκολύνουμε κιόλα ε, και την εφαρμογή και προώθηση αυτής της αρχής της νομιμότητας. Τελευταίο στοιχείο για το ADR, αν θα είναι δεσμευτικές ή όχι αυτές οι αποφάσεις. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποκατέσε με σαφήνεια, δεν έδωσε σαφείς κατευθυντήρες γραμμές επ' αυτού. Είναι όμως ένα θεμελιώδες στοιχείο αυτό. Αν οι αποφάσεις ενός σώματος ADR θα είναι δεσμευτικές ή όχι για τους καταναλωτές. Για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα του συστήματος ADR, οι αποφάσεις και η, έκβαση όσον αφορά τις αποφάσεις πρέπει να είναι δεσμευτική χαρακτήρα. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει δεσμευτικά να εφαρμόζονται υποχρεωτικά εκτός αν κάποιο από τα μέρη αποφασίσει να προσφύγει με δικαστικά σε σχέση με τα όσα είναι διαθέσιμα στα κράτη-μέλη. Αυτό που είναι σημαντικό είναι θα πρέπει να δραστηριοποιείται έτσι ο, ο, ένας ή ο άλλος ώστε να μην αγνοούνται οι αποφάσεις του ADR. Να μην δηλαδή ε, οδηγηθούμε στο να απεμποληθούν οι αποφάσεις αυτές. Τώρα, σε σχέση με μη δεσμευτικές ε, αποφάσεις, ε, ιδιαίτερα αν για κάποια κράτη έχει αποδειχθεί ότι αυτού του χαρακτήρα οι διαδικασίες ε, μπορούν να λειτουργήσουν στις σκανδιναβικές χώρες, παρότι τέτοιου είδους αποφάσεις μπορεί να μην είναι δεσμευτικού χαρακτήρα, μπορεί να, το σύστημα να λειτουργήσει μέσα σε τέτοια πλαίσια. Δεν έχω όμως χρόνο να υπησέθω σε όλα αυτά. Θέλω απλά και μόνο να απαντήσω στι ερωτήσει της κυρίας Τούν. Πιστεύουμε απόλυτα ότι το ευρώ θα πρέπει να είναι εθνικό αλλά και διασυνοριακού χαρακτήρα ε, διαφορών. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν θα πρέπει ο καταναλωτής να σκέφτεται θα αγοράσω σε ένα άλλο κράτος μέλος ε, ή στη δική μου χώρα ε, συνειδητοποιώντα αυτά. Είναι η εσωτερική αγορά πρέπει να δίνει την δυνατότητα οι άνθρωποι να μπορούν να κινηθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αυτό είναι σημαντικό. Το δεύτερο σημείο που αναφέρατε είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή ίσω είναι παραπλανητικό για του καταναλωτέ. Αν ακούνε μόνο για μία πλατφόρμα, λέει. Πρέπει να είναι μία πλατφόρμα ενημέρωση. Να κατανοούν οι καταναλωτέ ότι είναι για την ενημέρωση και πληροφόρησή του και όχι απλά και μόνο για μία διευθέτηση διαφορών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Πάκλη για μια πραγματικά πολύ περιεκτική και ε, χρήσιμη παρουσίαση παρά το ότι ξεπεράσατε λίγο το χρόνο σας. Από την Business Europe τώρα ο Πέντρο Ολιβιέρα ο οποίος είναι νομικός σύμβουλος από το 2009 και ασχολείται με ζητήματα δικαιωμάτων των καταναλωτών ε, και ε, ζητήματα αποζημίωσης. Άλλωστε έχετε και τα σχετικά στοιχεία του ε, στο φάκελό σας. Θα ήθελα να του δώσω το λόγο για να μας πει την άποψη της Business Europe για τις δύο αυτές προτάσεις. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της ε, ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, εμείς είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές των δύο αυτών προτάσεων, γιατί είναι ένας σύντομος και αποτελεσματικός, λίγο δαπανηρός τρόπος επίλυσης διαφορών, ε, εποφελής και για τους καταναλωτές αλλά και για τις εταιρείε. και είναι πολύ σημαντικό ε, να έχουν ε, άμεση πρόσβαση οι καταναλωτές σε αποζημίωση όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ε, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ε, συχνά οι καταναλωτές ε, διστάζουν να προβούν σε αγορές διασυνοριακές, γιατί δεν ξέρουν ακριβώς τι να κάνουν όταν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα, σε ποιον απευθυνθούν και υπό ποιες συνθήκες. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η εναλλακτική επίλυση διαφορών δίνει τη δυνατότητα αντιμετώπιση των ε, καταστάσεων αυτών. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό. Ένα παράδειγμα το οποίο προκύπτει από μια έκθεση των δικτύων, των ευρωπαϊκών δικτύων κέντρων καταναλωτών ε, ε, πώς λειτουργήσε το ADR στην, στην πράξη. Ένας Ιρλανδός καταναλωτής αγοράζει σε ένα γαλλικό website μία ε, φωτογραφική μηχανή και ε, μετά από ένα χρονικό διάστημα αποφασίζει να το στείλει πίσω. Ο Γάλλος έμπορος λέει ότι δεν θέλει να τον αποζημιώσει για το ποσό ε, γιατί έλαβε λέει πίσω ένα άδειο κουτί. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι μετά από επαφή του με τον έμπορο, ο καταναλωτής πήγε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών στη Γαλλία και ο έμπορος τελικά ε, επιβεβαίωσε ότι υπήρξε ένα πρόβλημα με, ε, τους, με, αριθμού, με, τα, με τους αριθμούς των πακέτων και τελικά έλαβα αποζημίωση. Ε, Slides don't move. <laughs> Ε, ε, θέλουμε να θεωρηθεί ένας από τους 12 μογλούς της ε, ε, ενιαίας αγοράς. Υπάρχουν βέβαια διάφοροι τρόποι τέτοιου είδους επίλυσης στην Ευρώπη και δεν υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να, ε, να υπάρχει κάτι τέτοιο γιατί δίνει την απαραίτητη, την απαραίτητη ευελιξία. Δεν είναι, δεν είναι τόσο το είδος ε, της εναλλακτική επίλυσης διαφορών, αλλά του να υπάρχουν αυτοί οι τρόποι επίλυσης διαφορών ε, να υπάρξουν εκεί που δεν υπάρχουν σήμερα και επίσης να επιφέρουν μια προστιθέμενη αξία. Ε, για παράδειγμα στο διαδίκτυο, ε, στο οποίο δεν υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι φορείς επίλυσης διαφορών εναλλακτικοί. Εμείς επικροτούμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα το γεγονός ότι υπάρχει ειδική πρόταση για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, το ODR, Υπάρχουν κάποιες ε, προσαρμογές που απαιτούνται και γι' αυτό θα αναφερθώ σε δύο-τρία σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι ένας, μία από τις βασικές ανησυχίες μας, ε, η ε, συνάδελφος από την Ένωση Καταναλωτών επίσης ε, το ανέφερε, άρθρο 2 παράγραφος 2α που αναφέρει ότι η οδηγία δεν θα ισχύει για τις διαδικασίες οι οποίες αντιμετωπίζονται από φορείς ADR αποκλειστικώς χρηματοδοτούμενοι από τον έμπορο. Αυτό το exclusively, το αποκλειστικά είναι που μας προβληματίζει. Εμείς ρωτάμε για ποιο λόγο, κατά την άποψή μας, αυτό το οποίο ε, διακυβεύεται εδώ δεν είναι τόσο η οικονομική ανεξαρτησία, αλλά η αμεροληψία. Για μας αυτό είναι το βασικό ζήτημα και σύμφωνα με άλλε ήδη υφιστάμενε οδηγίες ε, υπάρχουν κάποιοι σε ADR, να σα πω το παράδειγμα για παράδειγμα των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, ε, όπως επίσης ε, και του ασφαλιστικού τομέα και των χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Βλέπουμε ότι υπάρχουν λοιπόν πολλοί τέτοιου είδους φορείς στην πράξη που ήδη συμμορφώνονται με πολύ αυστηρούς κανόνες διαφάνειας. Για παράδειγμα, ε, τηλεπικοινωνίες ε, στη Γαλλία κάθε χρόνο εγκρίνουν μία έκθεση που παραθέτει τον αριθμό των ε, περιστατικών, πόσες υποθέσεις έπρεπε να αντιμετωπίσουν και προτείνουν μάλιστα και συγκεκριμένες συστάσεις στους ε, φορείς τηλεπικοινωνίας ε, για το πώς μπορούν να προσαρμόσουν τους όρους τους ε, για να είναι πιο συμβατοί με τον νόμο και η έκθεση αυτή υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλίας σε συλλόγους καταναλωτών και νομίζουμε ότι είναι πραγματικά ένα πολύ καλό παράδειγμα διαφάνειας. Άλλα παραδείγματα. Στη Γερμανία με τον ασφαλιστικό τομέα. Για μας το να μην τροποποιηθεί το άρθρο 2 ουσιαστικά αποκλεί ε, έναν μεγάλο αριθμό φορέων που είναι αμερόληπτοι και λειτουργούν εύρυθμα και δημιουργούν επιπλέον υποχρεώσεις στα κράτη-μέλη για ίδρυση νέων φορέων ADR ε, και εξέβρεση της νέας χρηματοδότητης σε περιόδους ε, κατά τις οποίες οι προπολογισμοί είναι πολύ περιορισμένοι. Πρέπει να είμαστε σαφείς. Αν τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να πληρώσουν, αν οι εταιρείε δεν πληρώσουν, ε, δεν υπάρχουν θαυματουργές λύσεις, ούτε μαγικές φόρμουλες. Αν λοιπόν ε, απαγορευτεί στους στον ιδιωτικό τομέα να χρηματοδοτήσουν τέτοιου είδους προσπάθεια, δεν θα βρεθούν ποτέ τα κονδύλια. Άλλη μας ανησυχία, το άρθρο 10, υποχρέωση ε, πληροφόρησης. Να αναφέρεται δηλαδή η πληροφόρηση για το ADR σε, οποιαδήποτε, σε κάθε απόδειξη και σε κάθε τιμολόγιο. Αυτό κατά τη γνώμη μας μπορεί να οδηγήσει σε λίγο βαριές καταστάσεις και νομίζω ότι μπορούμε να δείξουμε λίγο ρεαλισμό. Για μας είναι σημαντικό σαφής, ευ, σαφής εύληπτη αναφορά ε, στις φορείς ADR, είτε στον ιστότοπο, είτε στους όρους και προϋποθέσεις, αλλά νομίζουμε ότι αυτό είναι υπεραρκετό. Τώρα, επανερχόμενοι σε, σε κάποια από τα σημαντικότερα ζητήματα που εμείς ε, θεωρούμε ότι αναφέρονται στην οδηγία και είναι θετικά, δίνει το δικαίωμα ε, εθελοντικής ε, φύσεως για τους φορείς ADR. Αυτό είναι ένας από τους θεμέλιους λίθους του συστήματος και ενθαρρύνει ε, τη χρήση δικτύων ε, όπως ε, το, δίκτυο, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Καταναλωτών. Κάτι ακόμη, το οποίο ανέφεραν και οι δύο εισηγητές, για την ιεράρχηση της, ε, της αποζημίωσης κατά την επίλυση του προβλήματος. Συμφωνούμε καταρχάς ότι πρώτα ο καταναλωτής πρέπει να έρθει σε επαφή με τον έμπορο και φτάνω στο τέλος της παρουσίασής μου. Επίσης ε, θα ήθελα να είμαι και λίγο προκλητικός σε σχέση με τη συνάδελφο από το Σύλλογο Καταναλωτών. Εντάξει η ισότητα, αλλά η φορή ADR δεν είναι δικαστήριο. Μερικές φορές μπορεί να προσπαθούν βάσει ε, με δίκαιο τρόπο να προσπαθήσουν να επιλύσουν ένα πρόβλημα μεταξύ δύο μερών. Γιατί τα δικαστήρια είναι ακριβότερα και, εν πάση περιπτώσει, ε, αυτό που περιέγραψα περιμένουμε από τους φορούς ADR. Υποστηρίζουμε λοιπόν και τις δύο προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική και εναλλακτική επίλυση διαφορών. Ελπίζουμε ότι θα αλλάξει τη συμπεριφορά αλλά και τη στάση των καταναλωτών και των εμπόρων. Νομίζω ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις προτάσει αυτές και η Business Europe θέλει να είναι εταίρο στην προώθηση τη προσπάθεια αυτή ε, και στο να είναι τμήμα της εσωτερικής αγοράς ώστε να είναι μια προστιθέμενη αξία στην ε, ενίσχυση του διασυνοριακού εμπορίου. Ευχαριστώ. And, um, Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα πρέπει και ε, να υπάρχουν αντίτυπα αυτών που μας αναφέρατε. Να είμαστε σαφείς, ε, σίγουρα οι συνάδελφοι θα θέλουν να διατυπώσουν ερωτήματα όταν θα περάσουμε στον γύρο παρεμβάσεων. Τώρα, με ιδιαίτερη χαρά, θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Κορτές από την Ισπανία που είναι ε, στο Πανεπιστήμιο Λέστερ και έχει ευρύτατη πείρα σε σχέση με θέματα διαιτησίας και επίλυσης προβλημάτων ε, όσον αφορά θέματα καταναλωτών και έχει και διδακτορικό. Είσαστε ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος. Με ιδιαίτερη χαρά σας δίνω και εσάς τον λόγο για 8 λεπτά έχουμε νομίζω και στη διάθεσή μας εδώ θα πείτε. Θα έχουμε λοιπόν και με παρουσίαση με γραφήματα στις διαφάνειες. Έχετε τον λόγο κύριε Κορτές παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είναι χαρά για μένα να παρίσταμε σε αυτήν την ακρόαση. Θέλω να ξεκινήσω πρώτα συγχαίροντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σύνταξη και διατύπωση αυτών των προτάσεων από πλευρά της. Πιστεύω ότι ο ε, οδός προς το μέλλον είναι το ADR και το ODR, Alternative Online Dispute Resolution, για την επίλυση διαφορών. <clears throat> Είναι αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων, διευκολύνοντας την προσφυγή στη δικαιοσύνη στους καταναλωτές. Προσφυγή δυνατότητα να απονεμηθεί δικαιοσύνη για την επίλυση διαφορών, αντί να προσφύγουν σε δικαστήρια. Ξέρουμε ότι για τους περισσότερους δεν είναι αυτή η αυθεντική δυνατότητα να προσφύγουν σε δικαστήρια. Στα επόμενα λεπτά θα ήθελα να σας σκιαγραφίσω κάποιες προτάσεις ε, που θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε να έχουμε πιο αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των δύο εργαλείων, αυτών των δύο μέσων. Με την πρώτη πρόταση θέλω να προσθέσω την φωνή μου στους προλαλήσαντες που είπαν ότι πιστεύουν, όπως πιστεύω και εγώ, ότι η χρήση υπηρεσιών για τους καταναλωτές πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος σε τομείς που βρίσκονται υπορρύθμιση με συγκεκριμένο τρόπο να μπορεί κανείς να συμμετέχει. Θέλω να τονίσω τώρα τον όρο αποτελεσματικός για να υπάρχει συμμόρφωση με την αρχή της επικουρικότητας και την προσπάθεια επίλυσης διαφορών θα πρέπει το δυνατόν ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά να επιλύονται αυτές οι διαφορές. Θα πρέπει λοιπόν πρώτον να υπάρχει μια απέτηση να υπάρχει δυνατότητα με αποτελεσματικό προσπελάσιμο και προσιτό τρόπο όπου θα αυτό θα είναι διαθέσιμο. Και επίσης θα πρέπει να εντάσσονται και κάποιες διασφαλίσεις και εχέγγυα για εκείνους ε, τους ε, εμπλεκόμενους ε, και στις επιχειρήσεις που για παράδειγμα κανονικά δεν θα προέβλεπαν τέτοιες διευκολύνσεις από πλευρά επιχειρήσεων και εταιριών, αν υπάρχει μια υπηρεσία για τους καταναλωτές που δεν διαθέτει στοιχεία στη γλώσσα των καταναλωτών, τότε είναι σαφές ότι δεν πρέπει να επιλεγεί μια τέτοια διαδικασία εφόσον η γλώσσα δεν θα είναι κατανοητή. Ένα τρόπο λοιπόν να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδου καταστάσει θα ήταν να επιτρέπεται μια οπτικοακουστική πλατφόρμα να επιδεικνύει, να δείχνει στον καταναλωτή πού θα έπρεπε να βρουν δυνατότητα εφαρμογή αυτών των μηχανισμών οι καταναλωτέ. Οι πλατφόρμες αυτές πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από ε, τέτοιες μονάδες. Πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οπτικοακουστικές μονάδες, ε, audio platforms που θα δίνουν τη δυνατότητα και θα διευκολύνουν τα μέρη να, επιλύουν, να έρχονται σε επαφή και να επιλύουν τις διαφορές τους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνεται κάτι τέτοιο. Και μία δυνατότητα θα ήταν προφανώς να διευκολύνουμε και να δίνουμε στους καταναλωτές τις πληροφορίες που χρειάζονται κατά την ε, συγκυρία και στιγμή που έχουν κάποιο παράπονο και θέλουν να ασκήσουν προσφυγή. Κομμένες και ραμμένες πληροφορίες στις ανάγκες τους ε, για τους στόχους που θέλουν να, ε, να εξυπηρετήσουν, ώστε όταν υποβάλλεται ένα παράπονο από ένα καταναλωτή, θα εξαρτάται από αυτό το παράπονο ε, ποιε πληροφορίε θα του δίνονται για να μπορέσει να επιλύσει τι διαφορέ του, να επιτύχει την επίλυση διαφορών. Δεν θα πρέπει να ε, υπάρχουν επικαλύψει ε, στην προσπάθειά μα αυτή. Θα πρέπει ενώπιο ενωπίο να μπορούμε να προχωρούμε και με την δυνατότητα να ε, διαθέτουμε, για παράδειγμα, όσον αφορά τα κονδύλια, 400 ευρώ για επίλυση διαφορών, αυτό ε, σε σχέση με τα στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και έτσι με αυτόν τον τρόπο τίθενται κάποια πλαίσια, κάποια όρια. Θα πρέπει να διευκολύνουμε άμεσες λοιπόν διαπραγματεύσεις και άμεση επαφή και διευθέτηση των προβλημάτων μεταξύ των μερών μέσω αυτής της πλατφόρμας και της τεχνολογίας που προσφέρει. Μία άλλη δυνατότητα ως, προς, ως πρόταση είναι ότι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ε, δυνατότητες. Αυτό μπορεί να μην είναι αναγκαίο όταν μια επιχείρηση, μια εταιρεία έχει ήδη ένα τέτοιο, ε, μια τέτοια πλατφόρμα και έχει δεσμευθεί ότι μέσα από αυτήν θα δίνει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στα αιτήματα ή όπου η νομοθεσία ζητεί, απαιτεί από τους επιχειρηματίες ε, να είναι μέρος των συστημάτων ADR, Alternative ε, Dispute Resolution, ε, ώστε να μπορούν ε, μέσα σε αυτές τις διεργασίες, σε συγκεκριμένους τομείς, να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, εγχείρημα ADR. Επίσης θεωρούμε ότι είναι σημαντικό από την άλλη πλευρά να καταστεί σαφές στους καταναλωτές όπου και πού είναι αυτές οι υπηρεσίες διαθέσιμες στη γλώσσα τους. Οι επιχειρήσεις λοιπόν θα πρέπει να αποσαφηνίζουν αν το ADR προσφέρεται στη γλώσσα του ε, ετούντος ή στη γλώσσα του καταναλωτού. Τώρα, επίσης ε, θεωρώ ότι η ODR πλατφόρμα θα πρέπει online dispute resolution θα πρέπει και σε διασυνοριακές αλλά και σε εθνικές τέτοιες ε, επιλύσεις θα πρέπει να είναι μια εναλλακτική πρόσθετη δυνατότητα. Η πλατφόρμα ODR θα μπορούσε να χρησιμοποιείται ως αναπερίπτωση με εργαλείο διαχείρισης ε, και επίλυσης ε, προβλημάτων όταν υπάρχει ανάγκη να προσφύγουν οι καταναλωτές σε αυτό και να μπορούν έτσι οι επιχειρηματίες να βρίσκονται σε ένα σημείο κομβικό σε επαφή ώστε να μπορούν να έρχονται σε επαφή με αυτούς οι καταναλωτές από την αρχή ως το τέλος, χρησιμοποιώντας αυτή την εντό εισαγωγικών θηρίδα ή κομβικό σημείο, ώστε να μπορούν οι φορεί ODR να επικοινωνούν με τον καταναλωτή μέσω της πλατφόρμας ODR. Η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών είναι σημαντική υπόθεση και είναι εφικτή η δυνατότητα αυτή για τους καταναλωτές δεν θα πρέπει οι καταναλωτές να καταλήγουν σε μια άλλη δυνατότητα ή να προσφεύγουν σε άλλα μέσα πέρα από την ε, πλατφόρμα ODR από την αρχή ως το τέλος της διευθέτησης ενός παραπόνου που έχουν. Μια άλλη πρόταση θα ήταν και θα έλεγα ότι οι δεσμευτικέ, ή μη δεσμευτικέ ε, διεργασίε για τι ε, αποφάσει είναι δύο τελείω διαφορετικά πράγματα. Είναι πολύ διαφορετικά κότο το ένα από το άλλο, ιδιαίτερα όσον αφορά ένα συγκεκριμένο αριθμό ζητημάτων. Δύο θα ήθελα να αναφέρω τώρα. Πρώτον, το ότι πρέπει να αποσαφηνίσουμε αφενός υπό ποιες προϋποθέσεις και όρους ε, προδιαδικαστικές τέτοιες, προδιαιτητικές τέτοιες αποφα... Ε, διαδικασίες θα μπορούσαν να είναι δεσμευτικές ή όχι. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις στο ευρωπαϊκό δίκαιο γι' αυτό, αλλά δεν υπάρχει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο ή μια εναρμονισμένη εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι σωστό θα ήταν σε αυτό το σημείο να εξετάσουμε αυτή την πτυχή. Καθώς επίσης και σε δεσμευτικές τέτοιες αποφάσεις ή διεργασίες θα πρέπει να είναι δημόσια, δημοσιευμένο και διαθέσιμο το περιεχόμενο μιας τέτοιας απόφασης, ώστε μέσα σε μια διαφανή διαδικασία να γνωρίζουν όλοι το ποια απόφαση ελήφθη. Θα, ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην πυραμίδα αυτή που έχετε μπροστά σας στο γράφημα. Θα έπρεπε με άμεση ε, επικοινωνία μέσω της ODR πλατφόρμας να υπάρχει επαφή και στο τέλος τέλος μόνο ένα πολύ μικρό μέρος των ε, ε, προβλημάτων θα μπορούσαν να καταλήξουν στο επόμενο επίπεδο αν δεν έχει υπάρξει διευθέτηση προηγούμενα. Μια αποτελεσματική επίλυση αυτών των πρωτοβουλειών πρέπει να είναι σημαντικά κίνητρα για και τα δύο μέρη να συμμετέχουν και να, συμμετέχουν, να συμμετάσχουν στην επίλυση αυτών των διαφορών. Και τέλος πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία πάντα μεταξύ των πλατφορμών ODR, Online Dispute Resolution Platforms και των ε, κρατικών ε, ή επίσημων ε, δημόσιων αρχών ώστε να μπορεί να, ακολουθειται ακολουθείτε μια ταχύτατη διευθέτηση. Νομίζω η πλατφόρμα ODR θα ήταν το καλύτερο μέσο για να μπορέσουμε να ταυτοποιούμε ε, την, και να διασφαλίσουμε την συμμετοχή. Ξέρω ότι ξεπέρασα το χρονικό μου όριο, γι' αυτό ευχαριστώ για την προσοχή σας. Με ιδιαίτερη χαρά να απαντήσω σε ερωτήσεις αν υπάρχουν στη συνέχεια. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πράγματι πολύ για τα γραφήματα και τις διαφάνειες ε, που μας δείξατε, που ήταν, μας βοήθησαν πολύ. Τώρα θα ξεκινήσουμε λοιπόν ένα γύρο με ερωτήσεις και παρεμβάσεις από τους ομιλητές. Ανοίγει ο πίνακας εδώ για όσους θέλουν να συμμετάσχουν με αυτές τις ερωτήσεις από εσά. Ε, ε, ε, Η Κατιάνα Λαζότα, άρη νομικός από την Πολωνία και εργάστηκε και στην Ελβετία. Είναι εμπειρογνώμων σε, όσον αφορά νομικά θέματα που συνδέονται με το διαδίκτυο και πολλά από τα θέματα που άπτονται της ε, διαδικτυακής επίλυσης διαφορών και ADR συνδέονται όπως ακούσατε με την επίλυση ε, παραπώνων των ε, καταναλωτών από το διαδίκτυο. Κάτι που επαιδείει η Επιτροπή μας επί χρόνια όσον αφορά την ολοκλήρωση της ψηφιακής έννοιας αγοράς. Είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης της Ευρωπαϊκής για τα ψηφιακά μέσα. Οι εταιρείε δίνουν ψηφιακά προϊόντα στους καταναλωτές από το διαδίκτυο. Θα την καλέσω να μας δώσει τη δική της άποψη όσον αφορά την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ πολύ για την ωραία πρόσκληση να μπορέσω να έρθω εδώ να σας μιλήσω σε αυτό το πιο το επιφανές βήμα και θα ήθελα να αναφερθώ στην ένωσή μας. Στα μέλη μας έχουμε εταιρείε όπως eBay, Amazon και την εταιρεία που δουλεύω. Mm. Την MIH. Δεν λέει πιθανότατα πολλά για σας, αλλά έχουμε Είμαστε μέτοχοι σε διάφορες πλατφόρμες Κεντρική και Ανατολική Ευρώπης του διαδικτύου, οπότε θα μπορέσω να σας δώσω κάποιες ε, εικόνες, κάποιες ε, απόψεις για τους μεσάζους στο διαδίκτυο και το εμπόριο στο διαδίκτυο και το θέμα που συζητάμε. Είναι σημαντικότατο να εκφραστεί η άποψη των πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου και των μεσολαβητών στο διαδίκτυο, διότι είναι τα μεγαλύτερα βήματα όπου και τα δύο μέρη ε, συναντώνται, οι έμποροι και οι καταναλωτές, αυτοί τους οποίους συζητούμε, ε, ανεπτύχθησαν από τις ανάγκες και τα αιτήματα των καταναλωτών και το σημαντικότερο, πρόσφατες μελέτες που ετοίμασε η Copenhagen Economic έδειξε ότι οι μεσάζοντες του διαδικτύου συνέβαλαν περίπου στα 300, κατά 310 δισεκατομμύρια ε, ευρώ ε, στην ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι το μέγεθος της Ιλλανδικής οικονομίας. Θα σας δώσω άλλες πληροφορίες όχι τι γίνεται μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών μόνο, αλλά και τι ρόλο παίζουμε εμείς στην όλη διαδικασία. Θέλαμε, θα θέλαμε να υποστηρίξουμε τις πρωτοβουλίες αυτές ε, και είμαστε πεπισμένοι ότι θα συμμετέχουν, θα συνεισφέρουν στην εμπιστοσύνη ε, στην ευρωπαϊκή αγορά ε, και σίγουρα στην ανάπτυξη των διασυνοριακών συναλλαγών. Θα θέλαμε παρόλα αυτά να αποσαφινιστούν ορισμένα ζητήματα στη σημερινή συζήτηση. Αν εγώ βλέπω κάτι το οποίο είναι προφανές, ε, ε μπορείτε να με διακόψετε. Θα μιλήσω για ζητήματα τα οποία δεν είναι απολύτως ε, προφανή και κατανοητά για μένα όταν, όταν διάβασα το σχέδιο της, των προτάσεων. Ε, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι ε, ε, φυστάμενα, οι φυστάμενοι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών ε, που λειτουργούν μπορεί να μείνουν εκτός πεδίου εφαρμογής των προτάσεων γιατί υπάρχουν κάποιες εταιρείες που έχουν πολύ καλούς μηχανισμούς αντιμετώπισης τέτοιου προβλημάτων όπως για παράδειγμα η Amazon και θέλουν να συνεχίσουν ε, να λειτουργούν οι δικοί τους μηχανισμοί εφόσον υφίστανται. Θα ήθελα να σα επιστήσω την προσοχή σε ορισμένα νομικά ζητήματα. Είμαστε πεπισμένοι, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η ηλεκτρονική ενδιάμεση φορή ε, δεν θα ε, καλύπτονται από αυτές τις ε, προτάσεις. Δεν είμαστε έμποροι, δεν συμμετέχουμε στη σχέση εμπόρου και καταναλωτή και ο ορισμός ε, ηλεκτρονική παροχή αγαθών ε, και υπηρεσιών δεν είναι πολύ σαφής για μας. Σημαίνει μια συναλλαγή για την πώληση αγαθών, για την παροχή υπηρεσιών, όπου οι έμποροι προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες ε, ηλεκτρονικώς ή στον ιστότοπό τους και ο καταναλωτής έχει παραγγείλει με ηλεκτρονικό τρόπο ε, ή στον ιστότοπο τα αγαθά ή τις υπηρεσίες αυτές. Θα θυμάστε ε, Τώρα αυτό είναι τμήμα της οδηγίας ε, προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Πιο ήταν, ε, είχαμε νομίζω ε, κάποια προβλήματα πριν από τρία-τέσσερα χρόνια, τα οποία πέλησαν κάποια δικαστήρια στην Ευρώπη μπορεί ο κατανάλωτης, ε, έχει το δικαίωμα να ε, αποσυρθεί, να επαναχωρήσει μια, από μια αγορά και μας πήρε κάποια χρόνια ε, να το αποφασίσουμε αυτό και μέχρι σήμερα όντως έχει λυθεί το ζήτημα αυτό. Έχει τη δυνατότητα να επαναχωρήσει ο κατανάλωτης, να ασκήσει αυτό το δικαίωμά του αν ε, ε, δεν υπάρχει όμως αυτή η δυνατότητα, τότε ο καταναλωτής δεν έχει κανένα δικαίωμα επαναχώρηση. Εμείς θα θέλαμε να το αποσαφηνίσουμε αυτό, γιατί ακριβώς θα υπάρξουν για τα επόμενα χρόνια κάποια προβλήματα. Εμείς ε, ως ενδιάμεση στο διαδίκτυο θα θέλαμε να ξέρουμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Επίσης θα ήθελα να πω ότι θα θέλαμε να μην καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής των δύο αυτών προτάσεων. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πολύ ε, καλά προγράμματα προστασίας των καταναλωτών που εφαρμόζονται ήδη και δεν θα θέλαμε να υπάρχουν υποχρεώσεις για τους εμπόρους ε, που να ενημερώνουν, ε, να ότι δεν συμμετέχουν σε μια τέτοια εναλλακτική ή ηλεκτρονική επίλυση διαφορών γιατί αυτό θα έχει τελικά πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα των εμπόρων αυτών γιατί ένας έμπορος ο οποίος συμμετέχει στην όλη διαδικασία σε σχέση με κάποιον που δεν συμμετέχει, θεωρείται ότι ε, σέβεται περισσότερο τα δικαιώματα των καταναλωτών και ότι δίνει περισσότερα δικαιώματα στον καταναλωτή κλπ. Ε, θα ήθελα επίσης να θέσω και το θέμα το διασυνοριακό, το οποίο ε, ανέφερε και η Ούρσουλα στην αρχή. Για ποιο λόγο το ODR πρέπει να επικεντρώνεται μόνο σε, ηλεκτρο... σε ε, διασυνοριακές συναλλαγές. Μπορεί α πούμε να έχουμε μια τοπική πλατφόρμα από τι δικέ μας πλατφόρμες, Allegro, ενδεχομένως κάποιοι από εσά να τη γνωρίζετε, υπάρχει μόνο στην Πολωνία. Αυτή η πλατφόρμα αν δεν υπάρχει πίεση να οργανωθεί ένα φορέα ADR, ε, τότε θα έχει πολύ αρνητική εικόνα ε, και δεν θα υπάρχει κανένα τρόπο. Ε, για παράδειγμα, ο Πολωνό νομοθέτη δεν μπορεί να εισαγάγει ένα φορέα ADR χωρί να είναι υποχρεωμένο να το κάνει στο πλαίσιο τη οδηγία. Οπότε τέτοιου είδου πλατφόρμε μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Κάποια νομικά ζητήματα τώρα που θα ήθελα να θέσω. Όπως ενδεχομένως ε, να διαπιστώσατε, για τις δύο αυτές προτάσεις, στις δύο αυτές προτάσεις λέ, αναφέρεται ότι δεν θα, ότι θα πρέπει να ισχύουν δυνάμει του κανονισμού της Ρώμης όσον αφορά τις ε, συμβατικές ε, υποχρεώσεις και του, των Βρυξελών όσον αφορά ε, την δικαιοδοσία. Αν φτάσουμε σε μια εξή κατάσταση, ο καταναλωτή θα μπορούσε να έχει ενδεχομένως ε, υπό τον, ε, τους κανονισμούς αυτούς περισσότερη προστασία από ότι υπό, την, υπό τις προτάσεις, των προτάσεων που συζητάμε τώρα. Τι θα έπρεπε να κάνει. Θα έπρεπε υποχρεωτικά να δεχθεί την επίλυση σε επίπεδο ADR Υπτύχεται λοιπόν το θέμα του εφαρμοστέου δικαίου. Και επειδή περνάει η ώρα, θα προσπαθήσω να συνοψίσω. Αν υποθέσουμε ότι οι καταναλωτές συμφωνούν επί ενός αποτελέσματος, ποιο θα είναι αυτό. Αυτό ε, θα σημαίνει τι, ότι δεν πρέπει να ε, ξαναδικαστεί κάτι για το οποίο έχει ήδη υπάρξει δίκη ή κάποιο είδους, σε πάση περιπτώσει, αποκατάσταση ή ο έμπορος ε, πρέπει να γνωστοποιήσει στο φορέα ADR ε, μέσα σε 90 μέρες ε, τι έχει σκοπό να κάνει ε, ενώπιον του καταναλωτή. Ποια θα είναι η επιβολή τέλο πάντων τη όλη διαδικασία ώστε να εξασφαλίζεται το γεγονό ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών όντω προστατεύονται ε, σε τελική ανάλωση και ότι όντω υπάρχει ε, προστιθέμενη αξία από τι προτάσει αυτέ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Είμαι γενναιόδωρο στο χρόνο. Προσπαθούσαμε να βρούμε πού είναι η πολωνική διερμηνία. Εντάξει, τη βρήκαμε. Τώρα θα δώσω δυνατότητα να παρέμουν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή ε, Εσωτερικής Αγοράς που ασχολήθηκαν με αυτό. Ακούσατε από τους εισηγητές. Ε, θα ε, υπάρξει ανταπόκριση για θέμα να έρθουν στη συνέχεια. Οι σκιώδεις εισηγητές από τις κοινοβουλευτικές ομάδες εργάζονται από αυτής της πρότασης και άλλα μέλη. Ο κύριος Σουβάμπ λοιπόν που εκπροσωπεί τον κύριο Χάνς Πέτερ Μάιερ, σκιώδη εισηγητή για την πρόταση ADR, η κυρία Ρούλε, που είναι σκιώδη εισηγήτρια και για τις δύο προτάσεις, για την ομάδα των Πρασίνων, στη συνέχεια συνάδελφο από την ομάδα ECR. Έτσι λοιπόν νομίζω θα έπρεπε από αυτούς να ακούσουμε. Ο κύριος Μπαντασάρη θέλει να παρέμβει, ο κύριος Ρέπο επίσης ε, ο κύριος Ρέπο, ε, ε, αρμόδιος για την πρόταση ODR. Ας πάρουμε λοιπόν αυτό το γύρο ερωτήσεων, ξεκινώντας με τον κύριο Σουβάμπ, μετά στον κύριο Ρέπο, Ρούλε, Φόξ, Μπαλντασάρη και η κυρία Γκέπατ. Και μετά ο κύριος Γκράκ και η κυρία Τούν θα έχουν σίγουρα και εκείνοι κάτι να πούν. Ας πάρουμε αυτές τις παρεμβάσεις πρώτα και αυτές θα αναφερθούν στους εκπροσώπους ε, που θα έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν επ' αυτόν. Ο κύριος Σουβάμπε, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πραγματογνώμονες και ειδικού για τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Ήταν επικοδομητικό πιστεύω αυτό και για τις διαβουλεύσεις στις δικές μας επιτροπές και εργασίες. Γνωρίζουμε τους περισσότερους από τους συναδέλφους από τη διαβούλευση για την οδηγία για τα δικαιώματα καταναλωτών και δεν είναι τόσο διαφορετικά εδώ τα θέματα. Μια και έχουμε την ευκαιρία σήμερα τον συνάδελφο κύριο Μάιερ να τον εκπροσωπούμε στην οδηγία αυτή ε, για την ODR. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια θέματα που αφορούν την εκπρόσωπο της BOIC αλλά και τον εκπρόσωπο της Business Europe, τον κύριο Λιβέρα. Μπορώ να κατανοήσω καλά αυτά τα οποία είπε η κυρία Πάκλου ότι φυσικά μια βάση πρέπει να υπάρχει και να υφίσταται ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να βασίζονται στην νομιμότητα όσον αφορά τους καταναλωτές σε σχέση με το τι είναι διαθέσιμο για αυτούς στις χώρες τους. Αυτή πρέπει να είναι κάπως η αφετηρία για μια σωστή συμφωνία, για μια εξοδικαστική συμφωνία. Αυτός πρέπει να είναι ο πύχης, ο γνώμονας. Νομίζω είναι κάτι αυτονόητο αυτό και γι' αυτό ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το συμπεριέλαβε αυτό ρητά και κατηγορηματικά στο κείμενο της πρότασης προ την κυρία Πάχ και από τον συνάδελφο όπω μου το ανέφερε. Στο άρθρο 2, εδάφιο 2, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν περαιτέρω δυνατότητε και άλλοι τομεί που θα έπρεπε να ενταχθούν. Για παράδειγμα, όσον αφορά συμβάσει εργασία και απασχόληση. Τώρα, η συγκεκριμένη ερώτηση απευθύνεται και προ τον εκπρόσωπο τη Business Europe, τον κύριο Ολιβέηρα. Θα πρέπει να ενταχθούν ή όχι αυτέ οι πτυχέ. Δεύτερον, έχουμε το θέμα, το ζήτημα που απασχολεί τον συνάδελφο Μάιερ, το θέμα που αν σε σχέση με το κεφάλαιο 5 και το σκεπτικό 28, οι κυρώσεις και οι ποινές είναι κάτι επικοδομητικό ή όχι, πρόστιμα, ποινές. Και τι θα γίνεται πραγματικά στην πρακτική εφαρμογή στη συνέχεια. Θα μπορούσε ο ένα ή ο άλλο, η κυρία κυρια και ο κ. να απαντήσουν σε αυτό. Το τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι το θέμα τη υποχρέωση τη συμμετοχή δεσμευτικά σε τέτοιου είδου διεργασίε διευθέτηση διαφορών. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι ένα εθελοντικό σύστημα αν καταναλωτές θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό οι επιχειρήσεις. Αν όμως ξεκινάει η διαδικασία του ADR, η προσφυγή, οι αποφάσεις πρέπει να είναι δεσμευτικέ αν δεν υπάρχει προσφυγή σε δικαστήριο. Επ' αυτού θα μπορούσαν οι συνάδελφοι να πούν κάτι. Ευχαριστώ. Very much. Uh, Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ρέπο, παρακαλώ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τους, ε, τους για αυτές τις ε, εισηγήσεις από τη σκιώδη εισήγηση που έχω για τα θέματα ODR, αυτό το οποίο με ανησυχεί εμένα προσωπικά και είναι μέλημά μου, είναι να δούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την προσπελασιμότητα, την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για όλους, για τους καταναλωτές κυρίως, αλλά τους ευάλωτους καταναλωτές πάνω απ' όλα. Αυτό σίγουρα είναι και πρέπει να είναι κάτι που θα πρέπει να είναι ε, απλό και πρέπει να ρυθμιστεί. Ποιες δυνατότητες θα μπορούσαν λοιπόν να υπάρχουν και είναι δεδομένες για να πετύχουμε μια τέτοια υπηρεσία. Τέτοιου είδους υπηρεσία όπου θα μπορούσε να υπάρχει υποστήριξη, μια υπηρεσία που θα παρέχει συνδρομή και υποστήριξη ή συμβουλές για τέτοιους, τέτοια άτομα δωρεάν συμβουλές ή υπηρεσίες ή τουλάχιστον με τις πιο προσιτές δυνατές τιμές, τις χαμηλότερες δυνατές τιμές. Ευχαριστώ. Um, Κυρία Ρούλε τώρα παρακαλώ. Τα περισσότερα προαναφέρθηκαν από τους προλαλήσαντες. Γι' αυτό μια πρακτικού χαρακτήρα ερώτηση που θα ήθελα να αναφέρω, που από την κυρία Τούν προήλθε επίσης το θέμα, πόσες πλατφόρμες θέλουμε να έχουμε ακόμα για αυτόν τον τομέα. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει να συνταχθεί μια μελέτη πόσες τέτοιες πλατφόρμες θα πρέπει να υπάρχουν προτού εγκριθεί η ύπαρξη νέων τέτοιων πλατφορμών. Το θέμα για τις πλατφόρμες είναι παρόμοιο, είναι το ίδιο. Έχουμε το θέμα ε, ότι υπερβολικά πολλά υπάρχουν ευρωπαϊκά. Έχουμε ίσως κάθε γενική διεύθυνση που θέλει να έχει μια τέτοια ξεχωριστή πρόσβαση και μια τέτοια ξεχωριστή πλατφόρμα. Αν αυτό είναι το ιδιαίτερα φιλικό για τους καταναλωτέ, το αμφιβάλλω. Και σε σχέση με αυτό το οποίο έχουμε συζητήσει, κυρία Πάχρελ, για την ε, online dispute resolution. Είπατε ότι μπορείτε να το βαφτίσετε, να το αποκαλέσετε και διαφορετικά. Εντάξει, αλλά και το πεδίο εφαρμογής είναι σχετική υπόθεση. Όταν ισχύει για διασυνοριακές υποθέσεις, τότε μάλλον θα είναι δύσκολο για τους καταναλωτές. Αν το διευρύνουμε όμως σαν πεδίο εφαρμογής και για του εθνικού τομεί. Διαρωτώ με την ίδια συζήτηση θα έχουμε πάλι που θα επαναληφθεί όπως αυτή που είχαμε για την έκθεση Schwab. Έχω κάποια προβλήματα από τη μια πλευρά. Έχουμε προσδοκίες που δημιουργούνται για τους πολίτες και μετά ίσως δεν υλοποιούνται αυτές οι προσδοκίες, δεν, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν και αναμένει κάτι ο καταναλωτής online όσον αφορά εκεί τη θέση που έχει την έδρα του. Ευχαριστώ. Uh, Mr. Fox. Ο κύριος uh, thank you, Chairman. Can I also... Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους προσκεκλημένους μας για, την, για τις παρουσιάσεις τους. Ε, θα ήθελα να τους ρωτήσω ποια είναι η άποψή τους ε, σε σχέση με τις διαφορές ε, τις οποίες ξεκινούν επιχειρήσεις κατά των καταναλωτών, αν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στη συγκεκριμένη πρόταση ή όχι. Θεωρούμε συνήθως ότι οι καταναλωτές καταγγέλουν συνήθως επιχειρηματίες κατά το 99% των περιπτώσεων όμως ε, το αντίστροφο θα μπορούσε να αφορά μια ε, διαφορά που προκύπτει λόγω πληρωμής, καταβολής πληρωμής, μη καταβολής μάλλον. Οποιοδήποτε όμως, ε, οποιοδήποτε εσωτερικός μηχανισμός μπορεί να υπάρχει σε μια εταιρεία θα έπρεπε να προηγείται ε, του φορέα ADR, γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ε, αν πρέπει να περάσει πρώτα κάποιος από έναν εσωτερικό κανονισμό μιας εταιρείας. Πάνω από ένας ε, προσκεκλημένος είπε ότι ε, επειδή οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, αποθαρρύνονται από τέτοιου είδους ε, αγορές. Και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η βάση αυτής της, αυτής της δήλωσης και πώς είστε βέβαιος ότι μια τέτοιου είδους επίλυση διαφορών μπορεί να αυξήσει το εμπόριο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, οι περισσότεροι καταναλωτέ όταν αγοράζουν κάτι από ένα βρετανικό ιστότοπο δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά του και τα ε, μαθαίνουν όταν υπάρχουν ένα πρόβλημα. Δεν λέει κανεί, Α, όχι, δεν θα αγοράσω τίποτε ηλεκτρονικά γιατί δεν γνωρίζω τα δικαιώματά μου. Και υποθέτω ότι ισχύει το ίδιο για όλου του ιστότοπου, όχι μόνο του βρετανικού. Και μου φαίνεται ότι το πιο πιθανό εμπόδιο για έναν βρετανό καταναλωτή, ο οποίο συναλλάσσεται με ένα ε, μη βρετανικό ιστότοπο, άνθρωπο νομίζω ότι είναι το γλωσσικό εμπόδιο. Λιγότερο από 1% των καταναλωτών της χώρας μου γνωρίζουν μια άλλη γλώσσα ώστε να μπορούν να χειριστούν έναν άλλο ιστότοπο. Ε, ε, ένα πράγμα είναι να παραγγείλει κανείς έναν καφέ κάπου και άλλο είναι να πρέπει να παραγγείλει κάποιος έναν ιστότοπο, ένα αγαθό ή μια υπηρεσία. Το πρόβλημα λοιπόν το βασικό νομίζω είναι το γλωσσικό. For asserting that... Αναρωτιέμαι λοιπόν ε, πώς ε, μας διαβεβαιώνεται ότι θα αυξήσει το εμπόριο, ε, το διασυνοριακό, μια τέτοιου είδους πρόταση. Ευχαριστώ. Good. Uh, now, um, Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μπαλτεσάρη και μετά η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέσω ένα ερώτημα γιατί εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής Λοιπόν, όσον αφορά το, αυτά που συζητούνται, που είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Είναι πολύ χρήσιμη η ακρόαση με τους εμπειρογνώμονε που ήδη απάντησαν, πιστεύω, στι αντιρρήσει όσον αφορά την παραβίαση της αρχής επικουρικότητας και στο Κοινοβούλιο των Κάτω και στην Bundesrat, η γερμανική. Ετέθη το θέμα. Η έλλειψη αναγκαιότητας να υπάρχει ένα νομοθετικό μέσο, διότι θα αρκούσε ένα μέσο ρύθμιση επιθελοντικής βάσος όμως το άλλο κατά πόσο είναι σκόπιμο αυτό το εργαλείο της εναλλακτική επίλυσης των διαφορών μπορεί να ισχύει μόνο για τις διεθνείς σχέσεις, τις διασυνοριακές σχέσεις. Δύο ερωτήσεις θα να θέσω. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την αλληλεκτική επίλυση των διαφορών, κατά πόσο θα έπρεπε να σέβεται τις παραδόσεις ε, που ήδη υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Ε, πάνω απ' όλα, οι διάφορες ισομερείς συμφιλιώσεις, όπου συμμετέχουν οι ενώσεις καταναλωτών, εκεί, πέρα από τις επιχειρήσεις, ε, συστήματα που ήδη λειτουργούν με πολύ επαρκή τρόπο σε κάποιες χώρες, ξεκινώντας από τη δική μου. Τώρα όσον αφορά τις ευθύνες, τις αρμοδιότητες που δίνουμε στα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να εγγυώνται την ποιότητα των διαμεσολαβητών, αυτών που ασχολούνται με την επίσης διαφορών, ε, που θα εγγυώνται επίσης την παρουσία μιας αρχής, που αυτό προϋποθέτει ένα θελοντικό σύστημα επιλύσεως. Εκεί δεν χρειάζεται να συμμετέχουν οι ενώσεις των διαφόρων κατηγοριών που ήδη έχουν εμπειρία σε αυτόν τον τομέα και που εκπροσωπούν καταναλωτές και, ε, και βιομηχανίες και πωλήσει. Όσον αφορά την ε, ODR, online επίλυση διαφορών, εάν ε, δεν μπορούμε να το επεκτείνουμε και στις αγορές offline, ας πούμε fax, τηλέφωνο, τις συναλλαγές που δεν γεννώνται από άμεση σχέση μεταξύ δύο συμβαλωμένων μερών θα έπρεπε να μένει εκτός αυτή η πτυχή των εμπορικών συναλλαγών. Αυτό αφήνει μια κάποια τρύπα στο συνολικό πλαίσιο για την προσπάθεια των ε, ε, ρυθμίσεως αυτών των συναλλαγών σε ε, διασυνοριακό επίπεδο. Ευχαριστώ. Σημαντικά αυτά που λέτε. Κυρία Γκέπχαρτ, κάτι θέλει να πει. Ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση που μόλις τώρα την σκέφτηκα μετά από όσα είπε ο κύριος Μπαλτασάρη. Τι γίνεται τώρα με τις διασυνοριακές αυτές διεργασίες. Πώς θα τις ορίσουμε. Αν ζω στο και περάσω στο Στρασβούργο, περάσω το Ρήνο, online πάω να αγοράσω κάτι στη Γαλλία, όμως με τα προϊόντα αυτά επιστρέφω στη Γερμανία. Τι συμβαίνει, διασυνοριακή συναλλαγή είναι αυτή υπό αυτόν τον όρο ή όχι είναι μια ερώτηση που ίσως πρέπει να αποσαφινιστεί και αυτή. Για μένα είναι διασυνοριακή αυτή η συναλλαγή. Μπορεί όμως να πει επιχείρηση δεν είναι διασυνοριακή επιχείρηση, μια και σας φέραμε στη Γαλλία και αγοράσατε στη Γαλλία είναι ίσως θέμα ορολογίας και όρου, προσδιορισμού. Τι συμβαίνει εδώ, πώς θα τα καθορίσουμε όλα αυτά από πλευράς ορισμών, γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση και δεν λέμε ότι πρέπει να εντάσσονται σε ένα κοινό πλαίσιο. Είναι και μια ερώτηση προς την κυρία Πάχλ. Η δεύτερη ερώτηση που έχω είναι, και αυτή ήδη προαναφέρθηκε, είναι το θέμα των πλατφορμών. Νομίζω η κυρία Ρούιλερ το ανέφερε αυτό. Πόσες πλατφόρμες ακόμα χρειαζόμαστε. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν θα έπρεπε να σκεφτούμε ίσως μήπως αν υφιστάμενα όργανα ή φορείς, ίσως αυτή είναι η λάθος λέξη, ίσως υπηρεσίες που έχουμε και όργανα που έχουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για αυτό το σκοπό με τέτοιες αρμοδιότητες. Έχω υπόψη το κέντρο καταναλωτών, έχω υπόψη τα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών και άλλου φορεί Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ίσως αυτό θα ήταν μια απάντηση στην κυρία Ρούιλε στο ερώτημά τη. Γιατί και εγώ πιστεύω, όπως εκείνη, ότι όσο περισσότεροι φορεί και υπηρεσίε δημιουργούνται, τόσο πιο δύσκολο είναι οι καταναλωτές να βρούνε το σωστό δρόμο τι να κάνουν και δεν ξέρουν σε ποιον να στραφούν για να δικαιωθούν. Το τρίτο σημείο, για σε σχέση με ε, την προλαλή σα που ε, διαφωνεί ότι θα πρέπει να υποχρεώνονται, λέει, επιχειρήσεις σε μια τέτοια διαιτησία να συμμετέχουν υποχρεωτικά με το επιχείρημα ότι όταν αρνούνται θα έχουν κακή φήμη, λέει. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Θα μπορούσατε να μας τα επεξηγήσετε ακριβώς τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά, κυρία Λασότα, στην κυρία Λασότα το αναφέρω αυτό, όταν δουλεύει καλά μια επιχείρηση και σωστά αντιμετωπίζει τους πολίτες δεν έχει κανονικά κανένα πρόβλημα. Προβλήματα υπάρχουν μόνο εκεί όπου υπάρχουν προβλήματα από επιχειρήσεις. <laughs> Και γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω κυρία Λασότα, γιατί υπάρχει αυτός ο μεγάλος φόβος, αυτή η φοβία. Uh, ευχαριστώ. Θα επανέλθω στους δύο συγκητές μας που σημείωναν πυρετοδός, όπως και εγώ. Θα τους καλέσω να αναφερθούν σε κάποια σημεία και μετά θα επιστρέψω στο πάνελ για τυχόν σχόλια και κάποιες ε, απαντήσεις. Η κυρία Τούν πρώτα. Θα μιλήσω πολωνικά. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω πολωνικά. I wanted to give you the channel for um, Polish. Właśnie, właśnie, dobrze. Λοιπόν, ήθελα να έχετε, να βάλετε τα ακουστικά στο σωστό κανάλι για να ακούσετε. Ευχαριστώ πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Σε κοινό τώρα πάλι με τα πολωνικά για αυτή την συζήτηση, για αυτή την παρέμβαση. Είναι πραγματικά κάτι πολύ καλό να έχουμε αυτές τις αυτή την ενημέρωση σε σχέση με τις προτάσεις της Επιτροπής. Ε, πολλοί από εσά ανέφεραν ότι έχουμε αυτά τα διαφορετικά δίκτυα και σημεία σύνδεσης. Μπορούν να συνδεθούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους πολίτες όλα αυτά. Διότι υπάρχουν υφιστάμενες ενισχύ πλατφόρμες και η κυρία Ρούλε πολύ σωστά το κομψά το διατύπωσε. Οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για τις δικές τους, ας το πω δυνατότητες και στο τέλος τέλος μέσα από πολλές τέτοιες δυνατότητες χάνονται οι, χάνουν τον προσανατολισμό μέσα στο λαβύρινθο σε μια ας το πω έτσι ε, μεγάλη τέτοια ποικιλία δεν θα γνωρίζουν σε ποια θηρίδα ή σε ποια υπηρεσία να αποταθούν πιστεύω ότι όταν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει να είναι πιο εύκολο για τους καταναλωτές. Πρέπει να διευκολύνουμε στους καταναλωτές την πρόσβαση, την προσπελασιμότητα σε πληροφορίες εξ ου, άρα και για το δεύτερο ενημερωτικό έγγραφο και για, συμφωνώ με την κυρία Γκέπαρτ, δεν θα έπρεπε να διαιρούμε σε αλλοδαπής και ημεδαπής ε, υποθέσεις. Αναφέρατε κάτι, κάποια συναλλαγή ή αγορά. Πολλά τέτοια παραδείγματα μπορούμε να προσθέσουμε. Το πρόβλημα εδώ πολλές φορές είναι το γλωσσικό πρόσκομα, το γλωσσικό, ο γλωσσικός φραγμός. Από πλευράς Fox τέθηκε ένα ερώτημα σε σχέση με τη γλώσσα. Είναι σημαντικό αυτό. Τι θα κάνουμε, θα δημιουργήσουμε αυτή την νομοθεσία βραχυπρόθεσμα για σήμερα εδώ και τώρα ή για μακροπρόθεσμη χρήση. Ακόμα και σήμερα η χρήση τέτοιου είδους πλατφορμών για το διαδίκτυο το βρίσκουν οι καταναλωτές εύκολο να χρησιμοποιούν αγγλικά και είναι απλώς στις συναλλαγές τους. Δεν είναι πρόβλημα αυτό, αλλάζει ο κόσμος όμως και καμιά φορά προσπαθεί να τρέξει κανείς πίσω από τις εξελίξεις και πολλές φορές είναι ανεδαφική και παροχημένη η νομοθεσία και πρέπει να επικαιροποιείται. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε όχι το σήμερα, αλλά το αύριο το απότερο μέλλον. Και όσον αφορά τη γλώσσα, πιθανότατα αγγλικά. Αγγλικά θα είναι το πιο εύκολο να χρησιμοποιείται ως γλώσσα. Για προσφυγές αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα υστερότερα. Αν θέλει κάποιος να καταχωρήσει ή να οδηγηθεί σε διευθέτηση προσφυγής ή παραπόνου αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται στην γλώσσα καταχώρησης ή αποστολής του παραπόνου. Διότι αν έπρεπε να συνταχθεί σε μια ξένη γλώσσα αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα. Αν κάποιο είναι στο εξωτερικό ή όχι αυτό δεν είναι το κρίσιμο σημείο. Καμιά φορά χρησιμοποιεί κανεί μια πιστοτική κάρτα που έχει καταχωρηθεί στη χώρα του. Μετά πάει στο εξωτερικό, αγοράζει ένα προϊόν από μια τελείω ε, διαφορετική χώρα και μετά όταν βλέπουμε ότι γίνονται τέτοιες συναλλαγές, τι ακριβώς είναι διασυνοριακό πλέον σε ένα ευρύτερο τέτοιο πλαίσιο. Υπάρχουν λοιπόν θα έλεγα ασάφειες μετά. Δημιουργούμε κάτι για την, ως νομοθεσία για την παλαιότερη εποχή, για το χθες. Δεν ισχύουν όμως όλα αυτά πια σήμερα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε μια ενημέρωση, μια κρόαση για αυτά τα θέματα και να στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον. Προσέχοντας τις σημειώσεις μου, θα ήθελα να προσθέσω και ένα άλλο σημείο στα όσα προανέφερα. Ένα ακόμα. Ποιο είναι αυτό. Αυτό είναι το ότι ουσιαστικά πραγματικά ειλικρινά πιστεύω ότι δεν θέλουμε μόνο κάποιοι καταναλωτές. Φυσικά έχουμε πολλούς συναλλασσόμενους, έχουμε πολλές πλατφόρμες ε, σε σχέση με τις συναλλαγές online ηλεκτρονικά και υπάρχουν ε, ίσως ε, πολλοί πολιτές, αυτό ανέφερε η κυρία Λασότα, που έχουν μεγάλες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση καταναλωτών. Αυτό όμως που θα ήθελα να πετύχουμε είναι, προτού καταλήξουμε, προτού καταλήξουμε σε διαφορετικές νέες υπηρεσίες online θα πρέπει να κάνουμε κάτι απλό. Δηλαδή να έρθουμε σε επαφή πρώτα με τις επιχειρήσεις. Αυτή θα πρέπει να είναι η πρώτη επαφή με τον επιχειρηματή την επιχείρηση που μας πώλησε κάτι και ε, είχαμε συναλλαγή μαζί τους. Ε, λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνουμε. Να ενθαρρύνουμε τους καταναλωτές να έρθουν σε επαφή με τον εμπορευόμενο με τον οποίο είχαν κάποια συναλλαγή. Αν αποτύχει αυτό τότε υπάρχει το σύστημα ADR, Alternative ε, Dispute Resolution, να μην βρεθεί σε μειονεκτική θέση ο καταναλωτής, να μεριμνήσουμε, να διασφαλίσουμε ότι ο καταναλωτής θα μπορεί να διεκδικήσει και να διασφαλίσει τα δικαιώματά του στη γλώσσα του. Όμως πιστεύω ότι το έγγραφο θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ε, πτυχή του να υπάρχει εμπιστοσύνη, να υπάρχει δυνατότητα να στρέφεται κανείς προς τους επιχειρηματίες της επιχειρήσεις. Αυτό είναι σημαντικό, αυτό πρέπει να γίνεται. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μία ομάδα ενδεχομένων προβλημάτων είναι, αφορούν τον ορισμό. Τον ορισμό του δεσχυνοριακού, τον ορισμό του εμπόρου, τον μεσολαβητή στο διαδίκτυο, τον... εκεί θα πρέπει να δούμε τι είναι το ADR και λοιπά, τι είναι online και τι δεν είναι online, άρα θα πρέπει αυτό να το εξετάσουμε. Άλλος τομέας που νομίζω ότι αναφέρθηκε εκτενώς ήταν το θέμα των αρχών. Προφανώς έχουμε δύο αντίθετες απόψεις να αφορά τις αρχές της ανεξαρτησίας τι αποτελεί ανεξαρτησία. Αποκλειστικά απασχολούμενη, ε, νομιμότητα, τι είναι δεσμευτικό και τι δεν είναι δεσμευτικό. Τα πιο σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν περιεστρέφονται γύρω από τις τέσσερις αυτές αρχές. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση ήταν πώς μπορούμε να το επιβάλλουμε αυτό, να επιβάλλεται ο καταναλωτής. Εγώ θα έλεγα βασικά ότι θα ήταν και θέμα ε, δράσης μέσω δικαστηρίου, προσφυγή στο δικαστήριο. Εκπρόσωπος της Business Europe είπε ότι η αρχή της νομιμότητας συνεπιφέρει αυξημένη γραφειοκρατία και κόστος και θα έμοιαζε κάτι σαν κανονικό δικαστήριο και κάτι τέτοιο δεν θα λειτουργούσε. Θα ήθελα η, εκπρόσωπος από το ΒΕΟΚ να απαντήσει αυτό που είπε ο κύριος Ολιβέηρα. Θα ήθελα να ακούσω την απάντησή σας πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Ολιβέηρα. Θα με ενδιαφέρε. Σας ευχαριστώ. Καλώς. Θα στραφώ προς εμπειρογνώμονες σε λίγο. Ο κύριος Πιγκεντάλης ε, έχει κάτι να πει για τους εμπειρογνώμονες ως εισηγητή για την ΟΚΕΙΤ. Πάντα μου λένε ότι όταν υπάρχει η μητρική μου γλώσσα πρέπει να τη χρησιμοποιώ. Βλέπω ότι υπάρχει διερμηνία στα από πορτογαλικά. Θα μιλήσω πορτογαλικά, φορές τα ακουστικά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, λοιπόν. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι εδώ ε, θέλω να ευχαριστήσω για τις ε, προτάσεις και για τις ε, όσα αναφέρθηκαν και που θα υιοθετηθούν από πλευράς μας. Αυτά πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ή τρεις πτυχές, σε δύο ή τρία σημεία και να αναφέρω ποια είναι η θέση της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής όσον αφορά αυτές τις δύο προτάσεις που έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, σε σχέση με την πλατφόρμα ODR, Online Dispute Resolution εξέχοντα μέλη της Ευρωβουλής ήδη ρώτησαν πόσες τότιες λέει πλατφόρμες χρειαζόμαστε ακόμα εμείς. Ένα πράγμα είμαι βέβαιος ότι συμβαίνει. Αυτή την πλατφόρμα δεν τη χρειαζόμαστε σίγουρα. Δεν βοηθάει σε τίποτα αυτή η πλατφόρμα. Δεν είναι μια πλατφόρμα ODR αυτή όπως ε, από πλευρά συζητού αναφέρθηκε. Ο τίτλος ε, είναι παραπλανητικός. Αυτή η πλατφόρμα είναι αν θέλετε ένα πλαίσιο σαν ταχυδρομείο. Είναι ε, ένα σημείο όπου αποστέλλονται παράπονα και δίνουν, δίνονται απαντήσεις. Όλη η άλλη δουλειά γίνεται αλλού σε κανονικά γραφεία, κανονικά γραφεία επίλυσης ε, διαφορών σε κάθε χώρα μας. Και ήδη υπάρχουν αρκετά παραδείγματα πραγματικών πλατφορμών ε, για την επίλυση διαφορών ώστε θα έπρεπε να ε, υπάρξει καθορισμός ενός πλαισίου έτσι και όχι ενός ταχυδρομείου. Προσθέτω ακόμα παραπάνω σε αυτό ότι από τις γνώσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή η λειτουργία αυτών των αυθεντικών πλατφορμών ODR λειτουργούν καλά όσες υπάρχουν. Έχουμε αρκετά παραδείγματα από την Επιτροπή που θα μπορούσαν να έχουν παρακολου... α, ακολουθηθεί. Ίσως πρόκειται για ένα βήμα, ένα βήμα, πρώτο βήμα. Ίσως ε, υπό τους όρους αυτούς που έχει προσεγγιστεί το θέμα δεν είναι αναγκαίο. Τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν εδώ και οι ερωτήσεις που υπήρξαν για τις απαντήσεις που πρέπει να έχουν για τα θέματα γλώσσας, για τα θέματα cross-border ή μη cross-border, διασυνοριακών ή μη διασυνοριακών. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η πλατφόρμα για να είναι χρήσιμη δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις συναλλαγές online πρέπει να είναι σαφές ότι το πλαίσιο πρέπει να είναι διασυνοριακό για να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον αν υπάρχει ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, η γνωμοδότησή μας γι' αυτό ε, τοποθετείται η γνωμοδότησή μας για εναλλακτικέ λύσεις, επεξηγεί πρότυπα, θα τα βρείτε όλα αυτά στη γνωμοδότησή μας. Όσον αφορά το ADR, να πω ότι προφανώς ε, χαιρετίζουμε ως ε, Επιτροπή την μεταμόρφωση των συστάσεων soft law, ήπιας νομοθεσίας, σε οδηγία. Είναι προφανές αυτό. Αλλά έχουμε σημαντικές επιφυλάξεις όσον αφορά την χρήση από ε, επιχειρηματίες έναντι των καταναλωτών. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και επιφυλάξεις όσον αφορά τις ίδιες τις αρχές και τους προσδιορισμούς, τους ορισμούς. Υπάρχουν και οι συστάσεις ε, για, σε σχέση με την οδηγία που ε, έχασαν την ποιότητα του αρχικού ορισμού σε σχέση με την ε, αμεροληψία, την ανεξαρτησία και αμεροληψία που δεν είναι ακριβώς τα ίδια το ένα με το άλλο. Και μετά όσον αφορά και την φιλοδοξία, την φιλοδοξία αυτό το σύστημα να γίνει ένα γενικευμένο σύστημα που θα λειτουργεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σε όλες τις χώρες και σε όλες τις περιφέρειες και, ε, ε, περιοχές της Ευρώπης, ξεχνώντας το θέμα της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι θεμελιώδους σημασίας η διασφάλιση της χρηματοδότησης και ακόμα δεν έχει επιληθεί. Αλλά με ιδιαίτερο μεγάλο, τεράστιο ενδιαφέρον παρακολουθούμε την ε, τοποθέτηση επί της ουσίας της Επιτροπής ότι τέτοια συστήματα δεν υποκαθιστούν το δικαίωμα των καταναλωτών να προσφεύγουν στα δικαστήρια. Αυτή η αρχή που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τεράστια σημασία και μπορεί να ενισχυθεί βέβαια. Αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι το πρώτο βήμα, το πρώτο άνοιγμα που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τέτοιου είδους συστήματα για να μπορούν να εφαρμόζονται σε συλλογικές προσφυγές, σε ομαδικές προσφυγές ως ένα, ας το πω έτσι, πρώτο βήμα με την ε, ε, ελπίδα ότι αυτό θα δώσει την δυνατότητα να υπάρξει μια πραγματική αυθεντική συλλογική δράση σε, ευρωπαϊκή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα διασφαλίζεται έτσι. Εν πάση περίπτωση οι ευρωβουλευτές ήδη το ανέφεραν. Σε σχέση με τα σκεπτικά αυτής της πρότασης πρέπει να βελτιωθούν οι αιτιολογικές σκέψεις και να τις εκπονήσουμε με καλύτερο τρόπο στις νομοδοτήσεις μας αναφερόμαστε άρθρο προς άρθρο στις προτάσεις που κάνουμε για κάθε ένα από αυτά τα εδάφια. Αυτές οι επίση είναι διαθέσιμε στα αγγλικά. Αυτή η γνωμοδότηση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά στο site της Επιτροπής μας και θα εγκριθούν την επόμενη εβδομάδα και θα είναι στη διάθεσή σας από την επόμενη εβδομάδα και εφ' Ευχαριστώ. πάρα πολύ που ήρθατε και οι συγγητές θα το λάβουν αυτό υπόψη και ήρθε έγκαιρα η άποψή σας και θα θέλουμε να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτά που είπατε θα καλέσω την κυρία Ρουσό να σχολιάσει το τέλος. Ίσως θα ήθελα να ακούσει πρώτα την άποψη των εμπειρογνωμόνων και μετά θα τη δώσω και τη δυνατότητα να συνοψίσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα στραφώ προς του εμπειρογνώμονε τώρα, ακολουθώντας αντίστροφη σειρά. Ξεκινώντας από την κυρία Λαμότα, Λασότα, αν θα θέλατε να απαντήσετε σε κάποια από τα στοιχεία και τις ερωτήσεις που σας απευθύνθησαν για τις πτυχές online και αν είχα την καλοσύνη σε ένα δίλεπτο περίπου να καταφέρετε να απαντήσετε και να συνοψίσετε. Σας δώσω το λόγο λοιπόν να ξεκινήσετε εσείς. Να πω αυτό που είπε η κυρία Τούιν, ότι ανησυχούμε διότι πολλοί μπορεί έχουν ήδη καλά λειτουργούν τα συστήματα ε, και ίσως δημιουργηθούν πρόσθετα διοικητικά προβλήματα και βάρος εάν πρέπει να προσθεθούν πολλά ADR σε κάποιες χώρες όταν δεν ξέρουμε και πού θα βρίσκεται το ADR. Όταν επιλύονται προβλήματα καταναλωτών, όταν απευθύνονται σε εμά απευθεία. Δεύτερον, από ό,τι γνωρίζω, διαβάζοντας το κείμενο, εγώ θεωρώ ότι οι κανονισμοί είναι ήδη μη δεσμευτικοί, ότι είμαστε ελεύθεροι να συμμετάσχουμε στο ADR. Δεν είπα κάτι κατά του κειμένου. Απλώς ήθελα να είμαι σίγουρη ότι θα παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν και ήθελα να διευκρινιστεί ότι οι πλατφόρμες, οι μεσολαβητές στο διαδίκτυο είναι μεσολαβητές μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών. Και ότι δεν θα θεωρηθεί ότι εμείς ανήκουμε στο σύστημα ADR. Ας φανταστούμε λοιπόν ότι ασχολούμαστε εμείς με χιλιάδες εμπόρους, εκατομμύρια καταναλωτές και μετά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυξανόμενο αριθμό ADR ε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και ήδη πολλοί από εμά έχουμε ήδη ένα τέτοιο σύστημα ανάλογο. Οπότε ελπίζω αυτά που είπα να διευκρινίζουν την όλη κατάσταση. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Κόρτες έχει το λόγο. Δόκτωρ Κόρτες. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Συμφωνώ με το τελευταίο σχόλιο. Όπως αναφέρεται στον κανονισμό, είναι ODR η πλατφόρμα με την ενδεδειγμένη τεχνολογία. Το ADR να γίνει ODR ουσιαστικά με ενδεδειγμένη τεχνολογία. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της διευθέτησης μεταξύ των μερών όποτε είναι δυνατόν και θα πρέπει να διευθετεί τις περισσότερες διαφορές από την αρχή. Κάποιο στοιχείο να σας δώσω για το eBay. Το eBay πάνω από 60 εκατομμύρια διαφορές, ε, ε, διαφορές κάθε χρόνο διευθετεί. 60 εκατομμύρια το χρόνο. Γιατί και πώς. Αυτομάτως. Μέσω αυτόματων διαπραγματεύσεων. Η ομορφιά είναι ότι μοιάζουν πολύ οι διαφορές. Αγοράζουν κάτι online ε, φτάνουν καθυστερημένα τα εμπορεύματα και πολλά, πολλές διαφορές είναι παρόμοιες και οι διαμαρτυρίες είναι πολύ παρόμοιες. Όπως και τα διευθυντικά μέτρα είναι πολύ παρόμοια. Αυτό είναι το ωραίο. Να τονίσω αυτό που προανέφερα, ότι η πλατφόρμα θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, ούτως ώστε ο καταναλωτής να έχει στη διάθεσή του πληροφορίες και να διευκολύνεται και η διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των μερών. Στα γρήγορα, να αναφερθώ σε αυτό που προαναφέρθηκε. Κατά πόσο επιχειρήσεις θα μπορούσαν να έχουν αξιώσει έναντι των καταναλωτών όταν οι καταναλωτές δεν έχουν πληρώσει. Συνήθω, οι καταναλωτές πληρώνουν πριν πάρουν τα αγαθά. Ίσως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στην παροχή υπηρεσιών ή σε άλλε περιπτώσεις. Είναι σημαντικό να μπορεί να διευκρινιστεί σε ποιε περιστάσει θα, είναι, θα δεσμεύει και τον καταναλωτή μια συμφωνία εάν θα είναι αντίστροφη η σχέση. Σε ποιες ε, περιπτώσεις ο καταναλωτής θα είναι υποχρεωμένος να συμμετάσχει σε μια online διευθέτηση. Οι περισσότεροι καταναλωτές, αν τους ζητηθεί να συμμετάσχουν σαν ε, κατηγορούμενοι τους υπήρντες εισαγωγικών, δεν θα ε, συμμετάσχουν. Θα έχουμε πολλές περιπτώσεις που δεν θα πληρώνει καταναλωτής. Έχουν παραδείγματα πολλά στη ΣΥΠΑ που χρησιμοποιείται η διατησία επίλυση των διαφορών και δεν λαμβάνονται υπόψη όλες οι τυχές πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ολιβέρα έχει το λόγο. Νομίζω ότι ετέθησαν διάφορες ερωτήσεις που αφορούσαν εσάς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ολιβέρα, ευχαριστώ πρόεδρε. Ξεκινώντας με το θέμα το οποίο τέθηκε από τον κύριο Σουβάμπ, Πρώτη ερώτηση αν θα έπρεπε, αν υπάρχει ανάγκη να συμπεριληφθούν κάποιες άλλες περιπτώσεις εξαιρέσεων. Αντίστροφα θα το διατύπωνα. Ποιοι τομείς, ποια πεδία είναι εκείνα που πρέπει να προσπαθήσουμε να καλύψουμε, ποια πεδία για κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να μην καλύπτονται από το ADR. Το διατυπώνω διαφορετικά λοιπόν. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές συζητήσεις για κατόφλια, κατόφλια για αυτή την οδηγία μεταξύ άλλων. Αυτές οι ανησυχίες ε, θα πρέπει να μας κάνουν να λάβουμε υπόψη ακριβώς τη σαφήνεια που πρέπει να υπάρχει για τα κατόφλια στο, στην οδηγία αυτή. Γιατί αν αρχίσουμε να συμπεριλαμβάνουμε εξαιρέσεις, τότε στο τέλος θα αποκλείονται και οι μικρότερες εμβέλειας περιπτώσεις που και αυτές είναι σημαντικό να καλύπτονται από τα EDR. Μετά, για να απαντήσω την πρώτη ερώτηση του κυρίου Φόξ. Δηλαδή, αν οι επιχειρήσει θα έπρεπε να επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις διεργασίε ADR. Δεν έχουμε κάποια δεδομένη καθοριστική θέση επ' αυτού. Όμως άσχετα, κάνοντας λόγο για αυτήν την οδηγία ή όχι, θα ήθελα να λάβουμε υπόψη την εξή σκέψη αληθεύει ότι πλημμυρίζουν τα δικαστήρια με περιπτώσεις απουσίας πληρωμών, καθυστέρησης πληρωμών κτλ. κτλ. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να επιληθούν αυτές οι περιπτώσεις από το να πλημμυρίζουν τα δικαστήρια από τέτοιο κατακλυσμό περιπτώσεων και να παίρνουν χρόνια να ρυθμιστούν. Αυτός ο προβληματισμός είναι σημαντικό θα έλεγα να ληφθεί υπόψη και στα πλαίσια αυτής της ακρόασης. Ο κύριος Φόξ επίσης διατύπωσε μια ερώτηση, α το πω έτσι, για μια πρώτη επαφή με το in-house complaint scheme. Εντάξει, όμως αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ένα πλήρους εμβέλειας ε, in-house σύστημα, αλλά τουλάχιστον ένα πρώτο σημείο επαφής που θα μπορούσε να ακολουθήσει, διότι αυτό είναι η κοινή λογική που θα έπρεπε να εμπνέει τους επιχειρηματίες, αυτό θα έπρεπε να γίνεται. Τώρα για το θέμα το γλωσσικό, φυσικά η γλώσσα εξακολουθεί να είναι ένας φραγμός και αυτό έχει εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί πολλές φορές, αλλά σε σχέση με την τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Ιανουαρίου υπάρχει κοινή συμφωνία και συνένεση ότι είναι απουσία εμπιστοσύνης γενικά στην όλη κατάσταση διαδικτυακά δεν αγοράζει κάτι ε, σε ένα κατάστημα όπου γνωρίζει κανείς ότι μετά από δύο μέρες θα πάει στον πολιτή και θα ζητήσει να διευθετηθεί η διαφορά. Είναι διαφορετικό σύστημα αγοράς, διαφορετικό σύστημα εμπιστοσύνης, κάτι καινούριο και άγνωστο. Και κάτι καινούριο και άγνωστο χρειάζεται χρόνος για να διευθετηθούν όλα αυτά. Για τον κύριο Μπαλτασάρη, φυσικά οι νομικές παραδόσεις πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη. Και αν γίνονται σεβαστές ε, κάποιες παραδόσεις των χωρών μας, και αν σεβαστούμε τα ποιοτικά κριτήρια τα οποία αντανακλώνται σε σχέση με την οδηγία, γιατί όχι τότε θα έπρεπε να, είναι, να ενθαρρύνεται, να χρησιμοποιείται αυτό και να παραμένει στο σύστημα ζωντανό στοιχείο. Τώρα, ορισμοί. Θέματα ορισμών αναφέρθηκαν από αρκετού ευρωβουλευτέ, μέλη αυτή τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Σίγουρα πρέπει να δούμε τα θέματα ορισμών τους ορισμούς για διασυνοριακά θέματα, τι είναι διασυνοριακό, τι όχι και για την ανεξαρτησία φυσικά, διότι υπάρχει διαφορά σε θέματα ερμηνεία όσον αφορά την ας το πω έτσι, ε, έγκριτη, έγκυρη ερμηνεία και το πεδίο εφαρμογής. Μετά, συγκεκριμένα θέματα από τον εισηγητή κύριο Γκρέκ. Το τι εννοούσα εγώ με την δική μου εισήγηση είναι ότι δεν είναι το κάθε ADR ίδιο με ένα άλλο. Κάθε ένα είναι διαφορετικό. Έχουμε διαιτησία, έχουμε επιδιαιτησία, διαμεσολάβηση. Καμιά φορά ο φορέας ADR δεν δίνει κάποια απόφαση, απλά προσφέρει την πλατφόρμα να έρθουν ενώπιο σε ενωπίο οι εμπλεκόμενοι, να έρθουν σε επαφή και να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μια διαιτησία απόφαση στο τέλο. Ο ρόλο του EDR είναι να διασφαλιστεί ότι η νομιμότητα θα προστατεύεται και θα διασφαλίζεται. Να μην κοροϊδεύεται, να μην παραπλανείται και απατάται ο καταναλωτή και τα δικαιώματά του να διασφαλίζονται. Και σίγουρα, όπω είπε ο κύριο Πεγκάντολη, αν δεν είναι ικανοποιημένο ο καταναλωτή, μπορεί πάντα να προσφεύγει σε δικαστήρια. Και αυτό το προνόμιο το οποίο έχει ω δικαιώμα δικαίωμα δεν, δεν μπορεί να του αφαιρεθεί. Ευχαριστώ. Um, thank you for Ευχαριστώ για αυτές τις άμεσες απαντήσεις που δώσατε. Και τώρα η κυρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις, πάρα πολλές ετέθησαν και εκ των προτέρων απολογούμε διότι δεν θα μπορούσα να καλύψω τα πάντα. Προσπάθησα να ομαδοποιήσω τις απαντήσεις κάπως ε, ανάλογα με τις ερωτήσεις και θα ξεκινήσω με την ερώτηση για την νομιμότητα που ήταν το πρώτο σχόλιο του κυρίου Σβάμπ και ήταν ερώτημα που τέθηκε από τον κύριο Γκρέκ. σε απάντηση στην Business Europe είπε το EDR δεν είναι σαν δικαστήριο και δεν θα πρέπει να το φορτώσουμε υπερβολικά. Η απάντηση σχετικά με αυτό είναι ότι είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να υπενθυμηθούμε, να θυμηθούμε ότι τον Οκτώβριο του 2013 όταν θα τεθεί σε ισχύ η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών τα κάτι μέλη, ελπίζουμε, θα είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου που θα γίνει στην προσέγγιση στο ουσιαστικό δίκαιο και εξετάσαμε το θέμα πολύ προσεκτικά και όπως είπε και ο κ. είδαμε ότι τα βασικά παράπονα των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο περίπου στα ίδια πράγματα είναι η δικαίωμα από τις παραγγελίας, η παράδοση και εγγυήσει. Και δύο από τα βασικά κεφάλαια θα εναρμονιστούν πολύ σύντομα ε, και είναι μόνο η αποζημιώση της εγγυήσεις και οι περίοδοι που εκκρεμούν. Ε, νομίζω όμως ότι θα είναι εφικτό μέσω των φορέων του ADR να είναι ενήμερα για τα, τις αποζημιώσεις για τον καταναλωτή και για τις πλατφόρμες και για τα δίκτυα. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν προβλήματα. Ξέρουμε κάποιες ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών ήδη ε, εφαρμόζουν την αρχή της νομιμότητας στην πράξη και λειτουργεί και είναι θεμελιώδης πυλώνας της εμπιστοσύνης για τον καταναλωτή. Ξέρει ο καταναλωτής ότι δεν βασιστεί στα πρότυπα που γνωρίζουν και αν θέλει να δημιουργήσει κανείς εμπιστοσύνη, ε, νομίζουμε ότι είναι κρισίμου σημασία σε αυτό το στοιχείο. Όσον αφορά τους ορισμούς, που ίσως είναι κάπως ασαφείς, ίσως χρειάζονται και άλλοι ορισμοί, εξαιρέσεις επίσης από τους ορισμούς, ίσως θα ήταν χρήσιμο να προσθέσουμε έναν ορισμό σχετικά με το τι συμβάσεις καλύπτονται, δηλαδή να το δούμε θετικά το θέμα και θα ήθελα σε σχέση με την εξαίρεση των εστερικών φορέων διαμαρτυριών και εκείνων των ατόμων που απασχολούνται αποκλειστικά από μια εταιρεία να διατηρηθεί αλλά μπορούμε να δεχθούμε την περίπτωση όπου υπάρχει κάποιος φορέας επιχειρήσεων ε, και ε, απασχολεί κάποιον που ασχολείται με τη θέση των διαφορών. Και οι Ρώσοι σε τη λογική σκέψη 28, ναι, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσει σε περίπτωση που οι έμποροι δεν ανταποκρίνονται στι προδιαγραφέ και δεν ανταποκρίνονται στι υποχρεώσει του. Και θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσει από το κάτω μέλο. Σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Λαζότα, εσωτερικές ε, οι υπηρεσίε εσωτερικέ όπω Amazon και eBay, εσωτερικέ υπηρεσίε διαφορών, κάνουν πολύ καλή δουλειά τώρα. Δεν θα αποκλειστούν από την πρόταση ADR, θα εξακολουθούν να υφίστανται και μπορούν να συνεχίσουν. Και συντομού, συμφωνούμε ότι είναι σημαντικό να θαρρύνουμε του καταναλωτέ πρώτα να στρέφονται προ μια εταιρεία, προ τον φορέα διευθύνση διαφορών τη εταιρεία. Αν η διαδικασία που έχει η εταιρεία είναι αποτελεσματική, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μετά τέθηκε ένα ερώτημα τον κύριο Φόξ σχετικά με το να μην επαναλαμβάνουμε αυτά που ήδη υπάρχουν. Προφανώς δεν έχουμε ADR στην Ευρώπη με τρόπο προσβάσιμο και ολιστικό, άρα το χρειαζόμαστε. Και το ερώτημα είναι τι στοιχεία έχετε που αυτό θα προωθήσει περισσότερο δυσυνορικές συναλλαγές. στη διαβεβαιώ ότι έχουμε πολλά στοιχεία και με τα χαρά σας σας δώσω τα στοιχεία από, από όλα τα μέλη μα και την εμπειρία του από καθημερινέ επαφέ με του καταναλωτέ, ξέρουμε ότι το πρόβλημα στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι το ουσιαστικό δίκαιο, αλλά η πρόσβαση στην αποζημίωση. Ανησυχούν ότι αν πάνε στο εξωτερικό δεν θα έχουν κάποιον προ τον οποίο να στραφούν σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Τόσο απλό. Και οι μελέτε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι αυτό είναι το πρόβλημα υπαριθμών ένα στι συναλλαγέ, τι ηλεκτρονικέ, τι διασυνοριακέ. Το ερώτημα τη κυρία Γκέπχαρτ είναι διασυνοριακό. Πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα. Βλέπουμε πολύ μεγάλη ασυνέπεια όσον αφορά την νομοθεσία την ισχύουσα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να το προσεγγίσουμε το θέμα από την πλευρά των αποτελεσμάτων. Τι χρειάζονται οι καταναλωτέ, και πράγματι ένα Γερμανό καταναλωτή που ψωνίζει στη Γαλλία και περνάει τα σύνορα και είναι εκεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε ένα σύστημα EDR το οποίο είναι αποτελεσματικό και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να εστιαζόμαστε επί διαχωρισμού, να έχουμε ένα σύστημα το οποίο καλύπτει και τις διασυνοριακές συναλλαγές και τις εσωτερικές συναλλαγές. Αυτό θα λέγαμε και στην κυρία Ρούλε σε σχέση με το ερώτημα για την ενιαία πλατφόρμα. Γιατί να έχουμε και άλλη πλατφόρμα, δεν συμφωνώ με τον κύριο Πεκάδολης Έχουμε το Solvit, προφανώς υπάρχει, αλλά είναι πολύ διαφορετική πλατφόρμα, ασχολείται με πολλά διαφορετικά ζητήματα, όχι συγκεκριμένα ειδικά ε, με τις διαμαρτυρίες του, των καταναλωτών και την αποζημίωση των καταναλωτών. Χρειαζόμαστε κάτι ξεχωριστό, αποτελεσματικό, με συγκεκριμένο στόχο, να βοηθήσουμε τους καταναλωτέ. Δεν θα σε εκπλήσει ότι όσον αφορά κατά πόσο πρέπει να καλύπτει των επιχειρήσεων, εγώ θα έλεγα όχι, διότι είναι ένα μέσο που είναι συγκεκριμένο για την προστασία των καταναλωτών, οι επιχειρήσει είναι επιχειρήσει και έχουν άλλα μέσα στη διάθεσή του. Δεν είμαι σίγουρη αν κάλυψα τα πάντα, αλλά θα ήθελα να σταματήσω εδώ αν επιτρέπετε. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλώ, νομίζω ότι καλύψατε αρκετά θέματα, ευρύ φάσματα. Ευχαριστώ όλου σα πάρα πολύ για, το, για την ενθουσιώδη συμμετοχή σα και για τι σαφείς σα απαντήσει. Πρέπει να ολοκληρώσουμε στις 5, αλλά πριν το κάνουμε να δώσω στην Χριστίνα Ρουσό την ε, δυνατότητα να σχολιάσει τα όσα άκουσε σαν θεματοφύλακας ε, της προτάσεως και σαν ε, φορέας που έκανε, υπέβαλε την πρόταση. Χριστίνα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΙΝΚΟ και τους δύο εισηγητές που διοργάνωσαν αυτή την ακρόαση που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση Μόλις εχθέ ο πρόεδρος Μπαρόζο απέφθινε μια επιστολή στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων υπενθυμίζοντας την σημασία της έγκρισης αυτών των προτάσεων. Επίσης θέλω και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη προς την Δανέζικη Προεδρία του Συμβουλίου και για τα κράτη-μέλη που επιτελούν πολύ μεγάλο έργο για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι όπου όλοι και εμείς ως θεσμικά όργανα και ως ε, ε, εκπρόσωποι έχουμε συμφωνήσει να προχωρήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και για τις ε, παρεμβάσεις και την ευρεία υποστήριξη που εκφράστηκε για αυτές τις προτάσεις. Δεν θα έχω χρόνο τώρα για να απαντήσω σε όλες τις εξειδικευμένα τις ερωτήσεις σε λεπτομέρειες. Και σε σχέση με τις ερωτήσεις προς τους εισηγητές, πολλές ερωτήσεις απαντήθηκαν με καλό τρόπο από τα μέλη των εισηγητών, τους εκπροσώπους. Απλά και μόνο θα σχολιάσω κάποιες από τις πιο σημαντικές ε, παρεμβάσεις που έγιναν εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οδηγία EDR. Απόλυτα συμμεριζόμαστε τα σχόλια που έγιναν από τον εισηγητή κ. Γκρέκ που έχουν τεράστια σημασία αυτά τα θέματα, το εύρος αυτής της οδηγίας διασυνοριακά και εθνικά να διατηρηθεί και να διασφαλιστεί με πληροφόρηση και ενημέρωση των καταναλωτών που έχει τεράστια σημασία. Φυσικά θα πρέπει να συνδυάζουμε ένα ολόκληρο δίκτυο στοιχείων πληροφοριών για του καταναλωτέ, αλλά να μην αποτελεί αυτό υπερβάρηση, υπερβολική επιβάρηση για τι επιχειρήσει. Σημειώνουμε τις, ε, ε, τα, τα ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον που υπάρχει σε σχέση με του εμπλεκόμενου Για την αρχή τη ανεξαρτησία που αναφέρθηκε και από την Business Europe και από την BULK, Πιστεύουμε ότι από την Μπεκ, ήδη από το άρθρο 228 της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ADR καλύπτεται για την αρχή της νομιμότητας, μπορούμε να υποστηρίξουμε τη συμπερίληψη αυτής της αρχής, της ένταξης αυτής της αρχής στο κείμενο της οδηγίας. Όμως από την άλλη πλευρά φυσικά πρέπει να βρούμε μια διατύπωση σωστή που δεν θα επιβάλλει η υπερβολική επιβάρυνση δεν θα δημιουργεί ε, επιβάρυνση και εμπόδια στην λειτουργία του ADR. Ιδιαίτερα όταν βλέπουμε ότι προτείνουμε κάτι και δεν θέλουμε να το επιβάλλουμε διαβίας για το θέμα των ε, ε, εσωτερικών εκ των έσω internal systems για την αντιμετώπιση ε, προαραπώνων μπορούμε να υποστηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε τέτοιες δράσεις. Δεν μπορούμε όμως να υποχρεώσουμε τους καταναλωτές να ακολουθούν υποχρεωτικά μια τέτοια διεργασία διότι όλη η φιλοσοφική προσέγγιση αυτού του πακέτου είναι να χρησιμοποιούμε αυτά που υπάρχουν στα κράτη-μέλη και αυτά τα οποία είναι στη διάθεση του ADR. ADR και να αφήνεται ελαστικότητα, ευελιξία σε μεγάλο βαθμό, ώστε υπό τον όρο βέβαια πάντα ότι τα EDR θα συμμορφώνονται με τις ποιοτικές προδιαγραφές και διατάξεις ε, που είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα με αυτή την οδηγία, ο εφόσον θα εγκριθεί και θα ισχύουν αυτές οι διατάξεις μετά δεσμευτικά και για κάποια συγκεκριμένα σημεία στη συνέχεια για την ύπαρξη συγκεκριμένων περιπτώσεων ε, στα κράτη-μέλη ακόμα και όταν υπάρχουν σώματα διαιτησίας ε, που ασχολούνται με ε, αυτά τα θέματα, αυτό στο εδάφιο 6 ε, στην παράγραφο 6, στο άρθρο 6, εδάφιο 2 της οδηγίας καλύπτεται. Για συγκεκριμένα θέματα για το ODR, νομίζω πολλά από τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν λαμβάνονται υπόψη και σημειώνουμε φυσικά το γεγονός ότι υπάρχει, πώς να το πω, μια πολιτική, ας το πω, πολιτικού χαρακτήρα ζήτηση γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε διασυνοριακού ε, χαρακτήρα περιπτώσεις και τι πρέπει να θεωρείται διασυνοριακό σήμερα. Και στο σχέδιο κανονισμού παρέχουμε έναν ορισμό του TST διασυνοριακού χαρακτήρα για πιθανές τέτοιες διαφορές ε, στο άρθρο 4 Κατανοώ βέβαια ότι είναι ίσως νομικίστικη η απάντηση που σας δίνω επ' αυτού, όμως παρόλα αυτά είμαστε πολύ προσεκτικοί και ακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις συζητήσεις και τις εξελίξεις επ' αυτού του σημείου. Για μας ήταν ένας ορισμός, ένα περιορισμό στον ορισμό διασυνοριακά και να μην συμπεριλάβουμε τα πάντα. Και έτσι αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα που κάναμε πρώτο βήμα το οποίο αποφασίστηκε για τον ευδιάκριτο χαρακτήρα και τον ε, ας το πω έτσι διαρκέστερο πιο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα μακροπρόθεσμα και σε σχέση με τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να μπορούν από τους πόρους τους να παρέχουν δυνατότητες για τις διευκολύνσεις εκείνες που θα δίνουν τη δυνατότητα υποστήριξης αυτών των πλατφορμών. Όμως σημειώσαμε τα, διαφορετικά, τα διάφορα σχόλια που έγιναν και τις παρατηρήσεις και θα εισακουστούν πολύ προσεκτικά οι παρατηρήσεις των Ευρωβουλευτών. Και τώρα και φυσικά και ε, ως προς το Συμβούλιο. Φυσικά για το θέμα το οποίο αρκετές φορές αναφέρθηκε. Γιατί να υπάρξει ακόμα μια πλατφόρμα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούστε, δεν είναι ακόμα μια πλατφόρμα. Από ό,τι γνωρίζω φυσικά έχουμε συζητήσει και συζητούμε με όλους τους συναδέλφους. Δεν υπάρχουν άλλες πλατφόρμες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να αντιμετωπίζουν διασυνοριακά θέματα και θέματα συνδρομής για online επίλυση διαφορών σε σχέση με τις διασυνοριακές ή συναλλαγές ε, όσον αφορά επιχειρήσεις και καταναλωτές δεν είναι άλλη μία αλλά είναι ένα νέο μέσο αυτή η πλατφόρμα. Ένα μέσο το οποίο σαφώς θα έχει τη λειτουργία που περιγράφεται στον κανονισμό που προτείνουμε Ίσως θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη διατύπωση, θα μπορούσε να βελτιωθεί το κείμενο και οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται για τις λειτουργίες αυτής της πλατφόρμας και το σκοπό που εξυπηρετεί. Αν εγκριθεί ο κανονισμός ως έχει προταθεί, αν έστω και υπάρξει και κάποια τροποποίηση σε σχέση με το άρθρο 13 για παράδειγμα, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν πληροφόρηση πάντα και να υπάρχει άμεση προσπελασιμότητα και πρόσβαση σε αυτή την πλατφόρμα όταν έχουν κάποια συμβατική υποχρέωση που ε, ε, αναλαμβάνουν για, την, ε, κάποια συναλλαγή συμβατικά. Σημειώνουμε φυσικά τις παρατηρήσεις που έγιναν από την κυρία Τούν και άλλους ευρωβουλευτές αυτής της Επιτροπής και της Ευρωβουλής ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια διασύνδεση με τις άλλες ισχύουσες υφιστάμενες πλατφόρμες. Για παράδειγμα την ε, πλατφόρμα εκείνη που είναι εργαλείο και μέσο για τους Ευρωπαίους ε, πολίτες που πρέπει να δίνει δυνατότητα τέτοια διασύνδεση. Δεν υπάρχει πολλή χρόνο. Ολοκληρώνω εδώ. Ευχαριστώ για τη γόνιμη καρποφόρα συζήτηση και είμαι πρόθυμη να συνεχίσουμε υστερότερα με αυτέ τι επαφέ. Ευχαριστώ. Good. Um, Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Κριστίνα πάρα πολύ που ήρθες. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η ακρόση με συγκεκριμένο ξεκάθαρο στόχο. Πήραμε πολλές πληροφορίες, οι συγγητές θα πάνε και θα χωνέψουν πολλά από τα σημεία που εθίγησαν. Είπαμε ότι είναι πολύ αυστηρό το χρονοδιάγραμμα σε μία εβδομάδα να παραχθούν πρέπει εκθέσεις και νομίζω ότι μιλώ εκ μέρους και των δύο. Δεν νομίζω ότι είναι απόλυτα ε, έτοιμοι να κινηθούν πάνω σε αυτό, διότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία. Το όλο θέμα της ακροάσεως ήταν να δημιουργηθούν ερωτηματικά, να ακουστούν ερωτήσεις και να δοκιμαστούν κάποια από τα επιχειρήματά μας. Οπότε οι συντονιστές πιθανότατα αυτό σύντομα θα το συζητήσουν. Θα συζητήσουν ποιο θα είναι ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Θα έπρεπε να, παραδεχ... να λάβω υπόψη μου ότι είναι η κυρία Έλσκαρτ, ο, κύριος, η κυρία που, που προεδρεύει αυτόν τον είναι εκπρόσωπος της Δανέζικης Προεδρίας, αν θέλετε απλώς να παρουσιαστείτε, να συστηθείτε. Είναι πολύ καλό που είναι παρούσα η Δανέζικη Προεδρία, γιατί ενδιαφέρεται πολύ για το όλο θέμα. Λοιπόν, είστε πρόσδεκτοι να πείτε κάποια τελικά σχόλια. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι ήταν δύσκολη ημέρα για σας, εφορτωμένη και δεν θέλω να σας ε, κρατήσω εδώ παραπάνω. Ήθελα να σας πω ότι από την πλευρά, του Συμβουλίου θέλουμε, αναμένουμε εναγωνία συνεργασία ε, με ε, τους δύο εισηγητές για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα. δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά επ' αυτού και στο Συμβούλιο. με πολύ χαρά λοιπόν θα συνεργαστούμε με την Επιτροπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι η Δανική Προεδρία ε, δουλεύει πάρα πολύ σκληρά για τα ζητήματα των καταναλωτών. Την επόμενη, τον επόμενο μήνα μάλιστα ε, θα γίνει στη Δανία ε, στις 15 Μαρτίου στην Κοπενχάγη Παγκόσμια Μέρα Καταναλωτών. Ξέρω ότι ο κύριος Πεγκάντολής θα μεταβεί στην Κοπενχάγη γιατί η Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή συμμετέχει και εκείνη σε αυτά τα ζητήματα. Αν θέλετε να παραστείτε κι εσείς, ευχαρίστω να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ όλους. Ε, για τη συμμετοχή και τους προσκεκλημένους. Παρακαλώ να τους χειροκροτήσουμε. Uh, uh, Ελπίζω ότι θα συνεχίσετε να είστε σε επαφή με τους ε, εισηγητές μας ε, όσο συνεχίζουμε την προσπάθειά μας στο πλαίσιο των προτάσεων αυτών. Ευχαριστούμε επίσης και το ηλεκτρονικό μας κοινό, το κοινό που μας παρακολουθεί ηλεκτρονικός.